Ladies and gentlemen, please take your seats. Κυρίες και κύριοι, καθίστε. Κυρίες και κύριοι, καθίστε παρακαλώ. Good morning. Welcome everybody. In name of Mr. Καλώς ορίσατε εκ μέρους ε, του κυρίου Ομπερτφέλτ που θα έρθει σύντομα. Καλώς ορίσατε στην ακρόασή μας που έχει οργανωθεί υπό τον τίτλο «Ήδη πόρη και ε, και εναρμόνιση της φορολογικής ε, πολιτικής». Συνήθως ε, εδώ συζητάμε τα θέματα των δαπανών και όχι τόσο των εσόδων όμως, στο ευρύτερο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020 είναι καλό να πηγαίνουμε πέρα από τις γραμμές του προπολογισμού και να διερευνούμε το είναι ε, δυνατότητα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ε, ένα κύριο στοιχείο της συνολικής πολιτικής χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ξέρετε, μιλάμε για ένα περιορισμένο μόνο 2% είναι το ποσοστό που ανταποκρίνεται στις δημόσιες δαπάνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν αρκεί ε, για τη λειτουργία κλασικής σταθεροποίησης όπως έχουμε περνούν το στην περίπτωση του Ομοσπονδιακού Προπολογισμού των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρ' όλα αυτά έχουν εξεταστεί ήδη διπόροι από διάφορες οπτικές και ε, θέλουμε να αναζητήσουμε μετα... Ε, συνέργειες μεταξύ των φορολογικών πολιτικών ε, και των πολιτικών των κρατών μελών. Πρέπει να πω ότι βάσει της θεσμικής μου μνήμης ότι χρειαζόμαστε γι' αυτό ίδιους πόρους. Εδώ έχουμε ένα παράδοξο. Ε, δέχεται ε, κριτική το θέμα του ευρωπαϊκού προπολογισμού, όμως ε, εμένει. Και είχαμε βετεράνους αυτής της απόπειρας την τελευταία φορά. Ο κύριος Κάμερον ήταν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και ήταν πραγματικά αδύνατο να επιβάλλουμε το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ε, και να εναρμονίσουμε το ΦΠΑ. Τώρα ελπίζουμε με το Brexit να έχουμε ένα παράθυρο ευκαιρίας ε, να προχωρήσουμε και να σημειώσουμε πρόοδο στο θέμα των εσόδων. Θα έχουμε δύο πάνελ στην ακρόαση. Το πρώτο θα επικεντρωθεί στο πώς να συνδέσουμε καλύτερα τη φορολογική πολιτική και τις οικονομικές πολιτικές στην ενιαγορά αγορά και στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Το δεύτερο πάνελ αφορά τη φορολογική εναρμόνιση και το ε, δύσκολο θέμα του ε, να ε, μπορέσουμε τις κινητές φορολογικές βάσεις να τις συλλάβουμε μέσα σε εισαγωγικά. Έχουμε 20 λεπτά για τους ομιλητές και κατόπιν θα έχουμε ερωταπαντήσεις. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι έχουμε και αναμετάδοση στο διαδίκτυο της ακροασής μας. Εισαγωγικά θα έχουμε και δύο συνεισηγητές για τους ίδιους επόρους που θα πάρουν το λόγο. Θα δώσω το λόγο καταρχήν στην κυρία Βαλερή Αλιέ, η οποία είναι συνεισηγήτρια για το θέμα των ιδιών πόρων, για την εισαγωγή σας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να σας πω που χαίρομαι πολύ που οργανώνουμε αυτή την ακρόαση με τον Ζωζέ Μανουέλ Φερνάντες και θα συζητήσουμε του ίδιου πόρου. Είναι πολύ σημαντικό θέμα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επενθυμίσαμε σε ένα ψήφισμα του περασμένου Νοεμβρίου ότι δεν θα συμφωνήσουμε στο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο χωρίς να έχουμε πρόοδο στου ίδιου πόρου Και να είστε βέβαιοι ότι στο μήνυμα αυτό βρίσκει σύμφωνη όλη τη διαπραγματευτική ομάδα. Α μπούμε κατευθείαν στην ουσία. Η συζήτηση σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση του συστήματος ιδιών πόρων μας δείχνει το βαθμό υπευθυνότητας που θέλουμε να δώσουμε στην Ένωση και της εμπιστοσύνη που θέτουμε ε, σε αυτή. Ε, βέβαια, έχουμε μια ανησυχητική διαπίστωση. Δεν ε, έχουν μεταρρυθμίσει τα συστήματά τους τα κράτη από το 1998. Και όχι μόνο δεν έχει γίνει και μια μεταρρύθμιση εδώ και 30 χρόνια, αλλά το χειρότερο είναι ότι με την συμμετοχή σταδιακή αύξηση της ε, εθνικής ε, συνεισφοράς ε, και δεν ενισχύθηκε η συνεισφορά των κρατών μελών στον υπερεθνικό προϋπολογισμό. Αυτό θα μας ε, ε, ε, οδηγούσε σε μια ακραία κατάσταση. Φανταστείτε ότι βασιζόμαστε μόνο σε εθνικές συνεισφορές. Αυτό θα σήμαινε σαν να μην είχε έσοδο ένα κράτος μέσα από τη φορολόγηση των μισθών, χωρίς την φορολογική του πολιτική να την εστιάσει στην προστασία του περιβάλλοντος ή σε άλλες ενάρετες πρακτικές. Και θα αναφέρω ένα μόνο κράτος στον κόσμο που έχει μια τέτοια πολιτική. Δεν υπάρχει. Ε, και αυτό σχετίζεται με την αποδοχή του φόρου. Ε, έτσι όπως υπερασπίζει του ίδιους πόρους ε, το Κοινοβούλιο, οι ικανότητες που προσφέρονται από τον προπολογισμό μας είναι υπο, υποεκμετάλλευση σήμερα μου λένε να μιλήσω λίγο πιο αργά. Ε, το θέμα των εσόδων θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένα ξεχωριστό εργαλείο για να συνοδεύσει και να ε, συμπληρώσει τις ε, φορολογικές πολιτικές της Ένωσης. Έχουμε ένα απλό παράδειγμα, παραδείγματο χάρη, ε, τα έσοδα που προέρχονται από την κοινή ενωπημένη βάση φορολογίας των επιχειρήσεων, τι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για έσοδα όμως, ε, καταρχήν, θα μας βοηθούσε να καταπολεμήσουμε την ε, φοροδιαφυγή. Αυτό το περιμένουν οι Ευρωπαίοι. Ναι, ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών γιατί να θεσπιστεί για να καταπολεμήσουμε την κερδοσκοπία και για να προωθήσουμε περισσότερη φορολογική ισότητα. Είναι προσδοκία αυτή των πολιτών, ναι. Και ο φόρος ε, για τις ψηφιακές υπηρεσίες για να επιτρέψουμε να έχουμε καλύτερο διαχειρισμό των πτυχών ε, της ε, ψηφιακής εποχής, ε, ναι, είναι κάτι απαραίτητο και η συνεισφορά των πλαστικών ε, θα πρέπει να αποτελεί τμήμα της στρατηγικής της Κομισιόν για να μειώσει τα πλαστικά απόβλητα και να βελτιωθεί η ανακύκλωση. Και σίγουρα οι ωκεανοί θα είναι σε καλύτερη κατάσταση. Και φυσικά ο στόχος είναι ξεκάθαρος. Δεν θα πρέπει να εξφανιστούν αυτές οι αρχές. Στο μέλλον μπορούμε να εφαρμόσουμε τις ίδιες αρχές για άλλους τομείς δράσης της Ένωσης και ε, φυσικά το σύστημα εμπορίας ε, εκπομπών ε, και ο μηχανισμός προσαρμογή στα σύνορα μας βοηθούν να προστατεύσουμε το κλίμα. Πιστεύω λοιπόν ότι τα κράτη ποτέ δεν ήταν τόσο ανοιχτά ή θα έπρεπε να μιλήσω για ορισμένα κράτη-μέλη ότι ποτέ δεν ήταν τόσο κλειστά στο να έχουμε πράσινους πόρους. Έτσι λοιπόν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι και είναι ευτυχέ ότι και από καθαρά δημοσιονομική σκοπιά τα κράτη μόνο θα κερδίσουν να συστήσουν νέου ίδιου πόρου όχι μόνο θα φέρει αυτό έσοδα, αλλά θα μειωθεί και η εθνική συνεισφορά χρηματοδοτώντας τις δημόσιες ευρωπαϊκές πολιτικές ταυτόχρονα. Θα το καταλάβατε. Προτείνω το εξή. Από τη δεκαετία του 70, όπου είχαμε μια χρυσή εποχή για του ίδιου πόρους, έχασε δημοσιονομική πολιτική. Ε, συγγνώμη, δημοσιονομική αυτονομία η Ένωση. Και βρισκόμασταν μπροστά ε, στην βούληση των κρατών. Ε, όμως, ποια είναι τώρα η κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναμένεται φιλοδοξία και αποτελεσματικότητα για να απαντήσουμε στις προκλήσεις του 21ου αιώνα, προκλήσεις στις οποίες θα πρέπει ε, να απαντήσουμε και δεν γίνεται μόνο σε επίπεδο κρατών μελών. Και ε, θα πρέπει να έχουμε μια πολιτική γεωπολιτική Ευρώπη, η οποία προβάλλεται σήμερα από τη νέα Κομισιόν και από του αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων που κινητοποιούνται και από ένα νέο κοινοβούλιο που θα έχει τη δική του θέση στη διαδικασία. Είναι σε σημείο καμπή ε, η Ευρώπη και έχουμε και τη συνταγή να τη συνοδεύσουμε. Και σίγουρα η ικανότητα δράση τη Ευρώπη θα περάσει από θέσπιση νέων ίδιων πόρων. Ευχαριστώ όλου όσου είναι παρόντε εδώ και ελπίζω να διαφώτισα και τους ε, τελευταίους που δεν έχουν πιστεί για την αναγκαιότητα να έχουμε ένα νέο σύστημα ιδίων πόρων. Ευχαριστώ και τη Γραμματεία για την οργάνωση της ακρόασης αυτής ε, και Ζωζέ Μανουέλ, σου δίνω το λόγο. Thank you, Mrs. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Χαϊέρα για τα εισαγωγικά σας αυτά λόγια. Τώρα σας ακούσουμε και τον δεύτερο συνεισηγητή μας για τους ιδίους πόρους, τον κύριο Ζωζέ Μανουέλ Φερνάντες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και πράγματι χρειαζόμαστε αισιοδοξία. Θα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και ταυτόχρονα ρεαλιστές. Εγώ θα ήθελα να σας συγχαρώ και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλο το έργο που έχει υλοποιηθεί από τους εισηγητές του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την συνάδελφο, η εισηγήτρια Βαλερή, ε, για τη δέσμευσή της. Και ευχαριστώ και όλους τους προσκεκλημένους. Ευχαριστώ και τη Γραμματεία. Και μεταξύ των προσκεκλημένων θέλω να ευχαριστήσω τον Μιγέλ Πογιάρη Μαδούρο. Τώρα βρισκόμαστε σε ένα στάδιο που ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανταποκρίνεται είτε στις φιλοδοξίες των θεσμικών οργάνων, είτε στις προσδοκίες των πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει μια γεωπολιτική Ευρώπη, είναι αυτό προτεραιότητα της Προέδρου της Κομισιόν και γι' αυτό δεν μπορεί να έχει ένα προπολογισμό που να μην είναι επαρκής. Εμείς θα πρέπει να είμαστε το μοναδικό κοινοβούλιο παγκοσμίω που τοποθετείται επί των δαπανών και δεν τοποθετείται επί των εσόδων. Ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο να ε, υπάρξει, αναγκαιο... να υπάρξει ομοφωνία στο Συμβούλιο και κατόπιν υπάρχει έγκριση από κάθε Εθνικό Κοινοβούλιο. Όμως ε, ε, θα πρέπει να σεβαστούμε τις συνθήκες αλλά να αποφύγουμε ταυτόχρονα και την απλή επιστροφή του θέλω τα χρήματά μου πίσω. Αυτό για να μπορέσουμε να θεσπίσουμε πολιτικές προτεραιότητες πιο συγκεκριμένα και να ε, υλοποιήσουμε και τη Νέα Πράσινη Συμφωνία. Καθώς το Κοινοβούλιο δεν έχει δυνατότητα να γνωμοδοτήσει στο θέμα των ιδιών πόρων, εμείς ε, κάναμε κάτι που ήδη έχει λάβει η χώρα στο παρελθόν. Όμως θέλουμε να τονίσουμε ότι δεν ε, θα δώσουμε την εγκρισή μας στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο χωρίς ε, να υπάρξει μια νέα μεταρρύθμιση των ε, ιδιών πόρων. Εμείς θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια, θέλουμε να έχουμε ένα προϋπολογισμό που θα είναι ευανάγνωστος, θα είναι εύκολο να το κατανοήσει κανείς και ταυτόχρονα θέλουμε να μειώσουμε και το βάρος των εθνικών συνεισφορών και να έχουμε όμως και ένα επαρκές ποσό για να καλύψουμε τις φιλοδοξίες μας και ένα ρεαλιστικό ποσό για να το ένα 0,3% ε, ε, του καθάριστου χώρου εισοδήματο ανταποκρίνεται στην υλοποίηση των προγραμμάτων ε, και ουσιαστικά μα δείχνει και τι περιεχόμενο θέλουμε να δώσουμε σε αυτό το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Όταν μιλάμε για διευρυμένη μεταρρύθμιση του συστήματο των ιδιών πόρων, λέμε ότι ε, ναι, θα έχει νόημα για τα έσοδα από τα τελωνία, για τους τελωνικούς δεσμούς, το κάθε κράτος μέλος να κρατάει το ίδιο, το 20%. Επίσης, στην πολιτική ανταγωνισμού έχουμε τα έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως φυσικά είναι έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά κατόπιν πάνε στην τσέπη του κάθε κράτους μέλους μέσω διορθωτικών προπολογισμών. Είναι πιθανό να έχουμε μια απλοποίηση. Δεν έχει κανένα νόημα να έχουμε όλα αυτά τα rebates, όλες αυτές τις επιστροφές. Εμείς ε, θέλουμε να έχουμε πραγματικούς ίδιους πόρους. Στη φιλανδική πρόταση, το άνοιγμα, αυτή η δυνατότητα που δίνεται για να έχουμε νέους ε, ίδιους πόρους υπάρχει. Όμως ε, αυτό το άνοιγμα ε, έχει να κάνει με τη συνένεση για το θέμα των πλαστικών που έχει φυσικά και ένα θετικό σκοπό και αφορά τη συμπεριφορά του κάθε κράτους μέλους. Όμως, ε, ποιος είναι ο σκοπός εδώ. Αυτά τα έσοδα ε, τελικά να φτάσει στο 100% αν χρησιμοποιούνται όλα τα πλαστικά εκ νέου. Και δεν είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό το μόνο έσοδο από τα πλαστικά. Υπόθηκε ήδη και από τη συνάδελφο ε, έχουμε την ε, κοινή βάση φορολογίας των επιχειρήσεων. Θα μπορούσε να βοηθήσει αυτό το CCTB. CCCTB. Αυτό είναι ένα μήνυμα που θεωρώ πολύ σημαντικό. Ο δικός μας στόχος είναι να μειώσουμε, εάν μπορέσουμε, και την σωρά του κάθε πολίτη, όχι να ε, έχουμε νέα φορολόγηση των πολιτών. Να μην υπερφορολογούμε τους πολίτες και αν ε, πετύχουμε αυτή την εναρμόνιση μπορούμε να πετύχουμε εξοικονόμηση. Η Κομισιόν μας τα έχει αυτά, μας λέει ότι λόγω της φοροδιαφυγής και της ε, φοροαποφυγής χάνουμε πάρα πολλά χρήματα που αντιστοιχούν ε, ε, σε ένα προπολογισμό ευθετίας. Εμείς ε, θα θέλαμε να μειώσουμε το φορολογικό άχθος. Και εδώ τίθεται το θέμα της συνεισφοράς των μεγάλων ψηφιακών εταιριών δεν έχει κανένα νόημα οι εταιρείε ε, αυτές, ε, αυτές οι πολυεθνικές όπως ε, η Apple, το Facebook, η Amazon, η Google. Δεν έχει νόημα να μην πληρώνουν. Έτσι λοιπόν εμείς θα θέλαμε ακριβώς ε, να έχουμε και αυτή τη φορολόγηση για να μην υπερφορολογούμε τους πολίτες τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών επίσης είναι ένα ε, φόρος που θα έπρεπε να προωθήσουμε. Εμεί έχουμε την ε, δυνατότητα να εξυγχρονίσουμε τα έσοδα, να μπορέσουμε να καλύψουμε τους στόχους μας και ταυτόχρονα να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, καθώς θα έχουμε και το φόρο του άνθρακα στα σύνορα και να μπορέσουμε να αλλάξουμε τις συμπεριφορές και να συνδέσουμε αυτούς τους νέους ίδιους με νέους στόχους και αναφέρομαι συγκεκριμένα σε περιβαλλοντικούς στόχους. Έχουμε εδώ μεγάλη έμπνευση για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και ευχαριστώ εκ νέου τους προσκεκλημένους. Now... Σας ευχαριστούμε Ζωζέ. Ας περάσουμε τώρα στο πρώτο μας πάνελ, διασύνδεση της φορολογικής πολιτικής και του κοινοτικού προπολογισμού. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον φίλο μου Λάσλο Άντορ, που θα είναι ο πρώτος μας ομιλητής. Είναι γενικός γραμματέας του, Ιδρύματος, του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Προδευτικών Μελετών και από το 2010 στο 2014 ήταν ε, Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα απασχόλησης κοινωνικών υποθέσεων και ε, κοινωνική ένταξη. Είναι πλέον επιστημονικός ερευνητής στην Σχολή Διακυβέρνηση του Πανεπιστημίου του Βερολίνου, καθώς επίσης και επισκέπτης καθηγητής στο ULB, καθώς επίσης και στη Σιόν Σπο του Παρισιού. Μεταξύ 1991 και 2005, ο Άντοερ δίδαξε πολιτικές επιστήμες και οικονομική πολιτική στη Βουδαπέστη και ήταν, εκδότη ε, ήταν εκδότης μάλλον του προοδευτικού επιστημονικού περιοδικού «Εσμετελ». Επίσης συνέγραψε, δημοσίευσε δεκάδες βιβλία στην Ουγγαρία για ζητήματα οικονομικής πολιτικής, πολιτικής ιστορίας, συγκριτικών οικονομικών μελετών και για την παγκοσμιοποίηση. Το 2018 δημοσίευσε ο κύριος Σάντρο μια μελέτη με τίτλο πόροι για μια ευήμερη Ευρώπη, επανεσχεδιασμό του κοινωνικού προπολογισμού με έναν τρόπο προοδευτικό. Κύριε Άντορ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, για τα ευγενικά σας λόγια. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, χαίρομαι πάρα πολύ που επιστρέφω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμμετέχω στην συζήτηση αυτή. Συμφωνώ με του στόχου τη συζήτηση αυτή, να δούμε από οικονομική πλευρά πώ μπορούμε να μεταρρυθμίσουμε το σύστημα ιδίων πόρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και πώ μπορούμε να διερευνήσουμε νέου τρόπου βασιζόμενοι στη φορολογία για να έχουμε νέου ιδίου πόρου και πώ αυτό μπορεί να λειτουργήσει προ το συμφέρον των γενικότερων οικονομικών πολιτικών και των οικονομικών αποτελεσμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε φορά που συζητάμε ζητήματα δημοσιονομικά ή φορολογικά θα πρέπει καταρχάς να γνωρίζουμε τι θέλουμε να πετύχουμε με τα φορολογικά εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μα και πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε τα εργαλεία αυτά υπό το φω των στόχων που έχουμε θέσει. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θεωρώ ότι ε, κατέληξε σε αποτελέσματα η ψηλόβαθμη ομάδα εργασία του κυρίου Μάριο Μόντι μια υψηλόβαθμη ομάδα εργασίας η οποία υπέβαλε εξαιρετικές ιδέες βάσει μιας πολύ καλής ανάλυσης του τρόπου που λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και αναλύοντας βέβαια παράλληλα το εφιστάμενο τότε σύνολο εργαλείων. Εγώ θεωρώ ότι μια τέτοια ανάλυση όχι απλώς είναι δικαιολογημένη, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε κάτι ανάλογο με την έκθεση Μαγντούγκαλ του 1979 να καταφέρουμε να λύσουμε περισσότερο τις φορολογικές και δημοσιονομικές ικανότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σημερινή όμως εποχή. Θεωρώ ότι μια τέτοια ανάλυση θα ήταν δικαιολογημένη, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα χάσμα αξιοπιστία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ζήτημα αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τους Ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι αποφασίζουν να συμμετέχουν ή να μη συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές εκλογές. Το γεγονό ότι καταφέρνουμε και θέτουμε ω Ευρωπαϊκή Ένωση όλο και περισσότερου στόχου οι οποίοι συνδέονται με του πολίτε, είναι κάτι θετικό. Θα πρέπει όμω να γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ότι η φορολογική μα πολιτική και η φορολογική μα ικανότητα δεν είναι ενοποιημένη, δεν είναι πανευρωπαϊκή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε την πολιτική αυτή να τη διασυνδέσουμε με του στόχου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να καλύψουμε και να γεφυρώσουμε το χάσμα το οποίο υφίσταται αυτή τη στιγμή και το οποίο έχουν αντιληφθεί οι Ευρωπαίοι πολίτε. Στο πλαίσιο τώρα της υφιστάμενης συζήτησης βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ακόμα χάσμα, ένα χάσμα βιωσιμότητος. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή αν η φορολογική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι βιώσιμη και αν μπορεί να συμβάλλει στην δημοσιονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την οπτική λοιπόν αυτή γωνία θα πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί η φορολογική πολιτική. Ο Μόντι, ο Ζων Μπασιφέρη και άλλοι εμπειρογνώμονες τόνισαν κυρίω ότι υπάρχει μια λειτουργία κατανομής, διανομή του κοινοτικού προπολογισμού. Ακόμα και αν ο προπολογισμό αυτό είναι μικρός. Παρόλα αυτά καταφέρνει να συνεισφέρει πολύ σημαντικά στο να χρηματοδοτηθούν συγκεκριμένε ευρωπαϊκέ πολιτικές. Και αυτή, αν θέλετε, είναι και η βασική λειτουργία του κοινοτικού προπολογισμού. Και έχουμε και δύο βέβαια ακόμα λειτουργίες, την ανακατανομή καθώς επίσης και τη σταθεροποίηση. Ξέρουμε όμως ότι αυτή η ανακατανομή είναι αρκετά ασθενή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η λειτουργία της σταθεροποίηση ουσιαστικά δεν υφίσταται. Πρόκειται για ζητήματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν μόνο με την πτυχή των δαπανών, αλλά και με την πτυχή των εσόδων του κοινοτικού προπολογισμού. Τώρα, το αν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί με τρόπο βιώσιμο να συμβάλλει στη σύγκληση, την ευκταία αυτή σύγκληση, αυτό έχει να κάνει και με τις δύο αυτές πτυχές του κοινοτικού προπολογισμού. Έστω και δαπάνες, αν τελικά μπορούν να συμβάλλουν οι δύο αυτές πτυχές στον στόχο της αναδιανομής, της ανακατανομής. Και βέβαια αυτό εξαρτάται και από το μέγεθος του κοινοτικού προπολογισμού. Και από την οπτική αυτή γωνία μπορούμε να εξετάσουμε περισσότερο τα νέα εργαλεία τα οποία προτείνονται στην ε, νέα πρόταση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Τώρα, όσον αφορά την ασθενή λειτουργία σταθεροποίηση που έχει ο κοινοτικό προπολογισμό, ω προ αυτό θα πρέπει να εστιάσουμε λίγο περισσότερο στην πρόσφατη νομισματική μα πολιτική. Οι Ευρωπαίοι πολίτε, αλλά και άλλοι ενδεχομένω παράγοντε, ενδεχομένω να έχουν ανάμεικτα συναισθήματα όσον αφορά την νομισματική πολιτική που ακολουθείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι κάθε φορά που μιλάμε για προπολογισμό δεν αναφερόμαστε μόνο στον αριθμό των πόρων, γιατί εντάξει, αυτή είναι η βασική λειτουργία ενό προπολογισμού, να δώσει πόρου, αλλά θα πρέπει να δίδει επίση βασικού προσανατολισμού, καθώ επίση και κίνητρα. Θα πρέπει λοιπόν να φωτίσουμε και από αυτή την οπτική γωνία την όλη συζήτηση για τους ιδίους πόρους. Από ιστορικής πλευράς έχουμε δει στο παρελθόν ότι είχαν γίνει κάποιες προτάσεις στην περίοδο 2014 έως 2020 και κατά τη διάρκεια αυτού του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου έγινε μία πρόταση προκειμένου να έχουμε έναν φόρο επιχρηματοπιστωτικών συναλλαγών που αυτό όπως καταλαβαίνετε έχει να κάνει με συγκεκριμένα κίνητρα κίνητρα κυρίως θα δινόντουσαν από τον φόρο αυτό και όχι τόσο πολύ αυξημένα έσοδα ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα λειτουργούσε ω θετικό κίνητρο κατά των χρηματοπιστωτικών εκείνων συναλλαγών που δεν συνεισφέρουν και δεν ωφελούν, δεν ευνοούν την πραγματική οικονομία. Βέβαια, θα πρέπει, αν είναι εφαρμόσει κανείς ένα τέτοιο φόρο, να γνωρίζει και τι έστω θα μπορούσε να έχει από ένα τέτοιο φόρο. Ανάλογες ιδέες θα μπορούσαν να υποβληθούν προς συζήτηση. Για παράδειγμα, αν έχετε συγκεκριμένο στόχο πολιτικής, θα πρέπει να έχετε και συγκεκριμένα κίνητρα για την πτυχή των δαπανών ή για την πτυχή των εσόδων. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Εν είδη υποσημείωση, αν θέλετε, δεν λέω ότι θα κάνουμε αυτή τη στιγμή μια εκτεταμένη συζήτηση για το ζήτημα αυτό. Πάντω, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει μακροοικονομική σταθεροποίηση προσπαθεί να το πετύχει αυτό εδώ και πάρα πολύ καιρό, χωρί όμω να διαθέτει συγκεκριμένα εργαλεία πέρα από κάποιε συστάσει. Και γι' αυτό το λόγο αυτή τη στιγμή έχουμε πλεονάσματα στο ισοζύγιο συναλλαγών, τα οποία δεν έχουν μειωθεί, δεν έχουμε καταφέρει να τα μειώσουμε. Γιατί δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο εργαλείο το οποίο να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κράτη-μέλη τα οποία στον προπολογισμό του παρουσιάζουν πολύ μεγάλα πλεονάσματα θα ήταν πολύ σημαντικό αν μπορούσαμε να είχαμε ένα είδος φορολόγησης, ένα είδος εισφοράς, καταβολής ποσού που να επιβαρύνει τις χώρες εκείνες που παρουσιάζουν υπερβολικό πλεόνασμα. Στην περίπτωση αυτή, αν υπήρχε ένα τέτοιο εργαλείο, θα υπήρχε και ένα θετικό κίνητρο, προκειμένου οι χώρες αυτές να ακολουθήσουν συγκεκριμένε συστάσεις μετριασμού του πλεονάσματος. Κάτι άλλο, πέρα από τους πόρους και πέρα από τα κίνητρα θα πρέπει να δώσουμε και συγκεκριμένα μηνύματα ή αν θέλετε προσανατολισμούς ή κατευθυντήριες γραμμές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μπορείτε τουλάχιστον αν δέχετε τους απαραίτητους πόρους ή πολύ δυνατά κίνητρα να δώσετε κάποιους προσανατολισμούς όσον αφορά τουλάχιστον την πτυχή των δαπανών. Θα μπορούσατε για παράδειγμα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Πλάσα στο μέλλον να δώσει κανείς συγκεκριμένα κίνητρα όσον αφορά την κοινωνική συνοχή ή την κοινωνική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Αυτό ιδίω όσον αφορά την πτυχή των εσόδων και ιδίω όσον αφορά τον πολιτικό στόχο τη βιωσιμότητα. Ο στόχο αυτό τη βιωσιμότητα δεν αποτελεί βέβαια νέο στόχο στα πλαίσια του ορίζοντα 2020, ε, πριν από 10 χρόνια, όταν εκπονήθηκε η πρόταση αυτή, είχαμε ήδη μιλήσει από τότε για μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Πάντως, οι βασικές νέες ιδέες που είχαμε ακούσει κατά την προηγούμενη δεκαετία έχουν να κάνουν κυρίως με την πτυχή των δαπανών, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένε προϋποθέσεις, τη λεγόμενη ερεσιμότητα, προκειμένου να καταφέρουμε να πετύχουμε μια ευφυή βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμού. Θεωρώ ότι έχουμε εξαντλήσει πλέον τα όρια της πολιτικής αυτής και θα πρέπει να καταλάβουμε εκ νέου αυτή τη στιγμή για ποιο λόγο πρέπει να κινηθούμε περισσότερο προς την πτυχή των εσόδων. Δεν μπορούμε να θέσουμε περισσότερες προποθέσει. δεν μπορούμε να επιβαρύνουμε περισσότερο την αιρεσιμότητα όσον αφορά την πτυχή των δαπανών. Πρέπει λοιπόν να αρχίσουμε να μιλάμε όλο και περισσότερο για την πτυχή των εσόδων, πώ μπορούμε να αυξήσουμε τα έσοδα αυτά, πώ μπορούμε να δώσουμε κίνητρα μέσω τη πτυχή των εσόδων του κοινοτικού προπολογισμού. Και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι οι προτάσει Juncker και Entinger που γίνανε πριν από μερικά χρόνια είναι πολύ σημαντικό. Όσον αφορά την όλη συζήτηση για την επιστροφή, τα rebates στο πλαίσιο του προπολογισμού, νομίζω ότι είναι πλέον πολύ αργά για να ξεκινήσουμε τώρα μια συζήτηση η ε, επιστροφή που γίνεται ε, στο πλαίσιο του, της Βρετανικής συνεισφοράς είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να είχαμε ε, αντιμετωπίσει πολύ νωρίτερα. Το ίδιο σου αφορά και το φαινόμενο του grandfathering. Ζήτημα το οποίο θα έπρεπε να είχαμε αντιμετωπίσει πολύ νωρίτερα στα πλαίσια του κοινοτικού προπολογισμού. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν νέες, νέοι τρόποι που θα μπορούσαμε μέσω των οποίων θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της βιωσιμότητας του κοινοτικού προπολογισμού και των πεπερασμένων πόρων. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να δώσουμε κίνητρα ή να αντλήσουμε κάποια έσοδα από την φορολόγηση των μη ανακυκλώσιμων πλαστικών συσκευασιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι θέλει να προωθήσει ακόμα περισσότερο τους στόχους της βιωσιμότητας. Επί του παρόντο όμως φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αδυνατεί να μας πει από πού θα προέρθουν οι νέοι αυτοί πόροι που συνδέονται με τη βιωσιμότητα. Θα πρέπει να αποφύγουμε να χρηματοδοτήσουμε μέσω των εσόδων του κοινοτικού προπολογισμού την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία γιατί θα πρέπει να απευθυνθούμε μάλλον περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Τραπέζα Επενδύσεων ή σε άλλες δανειοδοτικές τράπεζες, προκειμένου να γίνουν οι επενδύσεις και να μην περάσουμε τόσο από φορολογία. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ήδη από πέρυσι ενέκρινε μια νέα στρατηγική και γίνεται μια ανάλογη προσπάθεια και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο πλαίσιο της νομισματικής της πολιτικής. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποφύγουμε την ε, όλη αυτή η προσέγγιση χρηματοδότησης Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας από τα έσοδα του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, τα κίνητρα που δίνει αυτή η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι πολύ σημαντικά. Ως προς αυτό, έχουν γίνει πολύ ενδιαφέρουσες προσπάθειες προκειμένου να καταφέρουμε να εντοπίσουμε νέες τρόπους χρηματοδότησης. Ένας αυστριακός οικονομικός επιστήμονας κατάφερε να εντοπίσει 7 διαφορετικούς τρόπους χρηματοδότησης του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ ότι οι ιδέες του αυτές θα πρέπει να κεντρήσουν το ενδιαφέρον μας, μολονότι ενδεχομένω να είναι πολύ αργά για να τις εφαρμόσουμε αυτή τη στιγμή. Η όλη επιχειρηματολογία μας που χρησιμοποιεί ο αυστηριακός αυτός επιστήμονας μπορούν να τροφοδοτήσουν, να εμπλουτίσουν τη συζήτηση που θα κάνουμε έκανε μια αναφορά, για παράδειγμα, ακόμα και σε ένα φόρο που θα βασίζεται στην πυρηνική ενέργεια ή στην διασυνοριακή καταβολή φόρου κάθε φορά που έχουμε μεταφορά πηγών άνθρακα και ούτω καθεξής. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχουν πολλές νέες ιδέες, πολλά νέα εργαλεία τα οποία θα μπορούσαμε να διερευνήσουμε περισσότερο για να ενισχύσουμε την πτυχή των εσόδων του ενωσιακού προπολογισμού και κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να δώσουμε και τα απαραίτητα κίνητρα για συγκεκριμένες εθνικές πολιτικές στα κράτη-μέλη. Και μία ακόμα πτυχή την οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι η ακόλουθη. Κάθε φορά που μιλάμε για έστω του προπολογισμού δεν μιλάμε μόνο για τον όγκο των εσόδων αυτών και για τα μέσα κίνητρα που δίνονται, αλλά και για το ζήτημα της διαφοροποίησης. Πώς μπορούμε να σταθεροποιήσουμε και να καταστήσουμε πιο βιώσιμο τον προπολογισμό. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να καταφέρουμε να διαφοροποιήσουμε τους σπόρους των εσόδων για λόγους βιωσιμότητος και αυτή η πτυχή θα πρέπει να αποτελέσει κέριο τμήμα της σημερινή μας συζήτησης αλλά και τη συζήτηση που θα κάνουμε στο μέλλον. Πρώτον λοιπόν να έχουμε το απαραίτητο ποσό στον νοσιακό προπολογισμό. Πραγματικά θέλουμε ο προπολογισμό αυτός να έχει καθοριστικό ρόλο στο δρόμο προς μία πιο βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς αποκλεισμούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσω προπολογισμού να δώσουμε θετικά κίνητρα. Θα πρέπει να αποφύγουμε οποιαδήποτε παράτυπη συμπεριφορά ή δεν θα πρέπει ο κοινοτικό ε, προπολογισμό ε, να χρηματοδοτεί λανθασμένε πολιτικέ. Διαφοροποίηση επίση των πόρων προκειμένου να καταστήσουμε πιο ανθεκτικό τον προπολογισμό μα και ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση αργά ή γρήγορα αναγκαστικά θα πρέπει να κινηθεί προ ένα συντονισμό των εθνικών φορολογικών πολιτικών. Αφού γίνει κάτι τέτοιο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε και την αρχή τη δικαιοσύνη, τη ισότιμη εφαρμογή ενό τέτοιου συντονισμού. Θα πρέπει ο ενωσιακό προπολογισμό να συμβάλλει στην ισοτιμία αυτή και να μειώνει τελικά τις ανισότητες που αυτή τη στιγμή φύστανται μεταξύ των κρατών μελών. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ Λάσλο. Και τώρα δεύτερος ομιλητής μας είναι ο καθηγητής ε, Μιγέλ Πογιάρης Μαδούρο από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο διευθυντής ε, της Σχολής ε, Διεθνικής Διακυβέρνησης με το 2009. Ήταν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο από το 2013 το 2015 ήταν αναπληρωτής, ε, μάλλον αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης Πρωτογαλία και γενικώ ε, έχει ε, διατελέσει σε πολλά αξιώματα σημαντικά. Έχετε το λόγο τώρα εσείς, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που με κάλεσε εκ νέου εδώ. Έχω έρθει αρκετές φορές Επίσης δεν είναι η πρώτη φορά που καλούμε να μιλήσω για τους ε, δύο σπόρους. Είναι ένα θέμα το οποίο εδώ και χρόνια συζητείται, το βλέπουμε. Βέβαια αυτό το ποτήρι εντό αγωγικών ε, μισογεμάτο ή μισοάδιο, εγώ προτιμώ να το βλέπω μισογεμάτο, διότι όταν προτάρισα να συζητώ για αυτό το θέμα, με θεωρούσαν σχεδόν τρελό. Κάτι που δεν ισχύει πια. Άρα, έχουμε λόγους να είμαστε πιο ε, αισιόδοξη. Δεν έχω πολύ χρόνο, θα ήθελα λοιπόν να εστιάσω σε δύο σημεία την παρέμβασή μου. Δύο σημεία που δεν συζητούνται ίσως τόσο πολύ ε, στο πλαίσιο των δύο πόρων. Και θα είπαμε λίγο με το Λάσλο πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση αυτή. Το πρώτο είναι ότι ο πρωταρχικός λόγος που είναι ανάγκη να επεκταθεί το σύστημα των ιδίων πόρων, κατά την άποψή μου δεν είναι οικονομικός, αλλά πολιτικός και έχει να κάνει με την νομιμοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και ε, σε επίπεδο εθνικών πολιτικών κοινωνικών. Η νομιμοποίηση εξαρτάται και από τον όγκο και από την ίσπραξη και την κατανομή διαφόρων πόρων. Ε, και αυτό είναι το βασικό μου σημείο. Το πρώτο. Το δεύτερο θα πραγματευθώ είναι σε ποιο βαθμό μπορούν τελικά ήδη οι πόροι επέκταση του συστήματο αυτού μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική ε, και πιο εφικτή εναλλακτική λύση ε, απέναντι στη φορολογική εναρμόνιση. Έχω κάνει προτάσεις ε, και σε μια έκθεσή μου που υπέβαλα το 2012 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το 2018 προσπάθησα να δοκιμάσω στην πράξη ε, στο, στη σχολή της ε, Διεθνικής Διακυβέρνησης, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο. Προσπάθησα λοιπόν να δοκιμάσω και είχα μια μελέτη με 10 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ε, πραγματεύτηκε διάφορα. Το πρώτο ήταν να μετρήσουμε ε, το βαθμό αλληλεγγύης που νιώθουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε υπηκόους άλλων κρατών της Ένωσης. Ε, τους ρωτήσαμε λοιπόν αν σας ενδιαφέρει το ίδιο, λιγότερο, εν μέρη κτλ. Και βλέπετε τα αποτελέσματα που ουσιαστικά είναι ισορροπημένα. Κάτι που αναμένεται είναι ότι οι περισσότεροι εν μέρη ενδιαφέρονται για τους πολίτες άλλων κρατών μελών, όχι το ίδιο δηλαδή με τα, ε, δεν τους νοιάζουν τόσο τα συμφέροντα άλλων όσο αυτά των συμπολιτών τους. Βλέπετε ε, τα πρόσφατος ε, προσχωρήσαν τα κράτη και τις χώρες του Νότου προς τα δεξιά και τα άλλα προς τα αριστερά. Το δεύτερο που θέλω να δείξω είναι μια άλλη ερώτηση. Τι προσδοκίες έχουν οι πολίτες για το τι μπορούν να αποκομίσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν υπήρχε ένα ταμείο λυγγύης μπορεί κανείς να συναγάγει πολλά συμπεράσματα. Εδώ βλέπουμε όμως ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συσχέτιση μεταξύ του βαθμού στον οποίο νιώθει κάποιος αλληλέγγυος και είναι ανοιχτό στην αλληλεγγύη ε, με το πόσα μπορεί ε, να θεωρεί ότι θα αποκομίσει από την Ένωση και οι άλλοι νοιάζονται δηλαδή. Η αλληλεγγύη έχει μεγάλη συσχέτιση με το τι θεωρούμε ότι θα αποκομίσουμε. Τι μπορούμε να περιμένουμε ότι θα κερδίσουμε από την αλληλεγγύη. Αυτή είναι μια γνωστή μεροληψία βέβαια. Ε, αλλά οι πολιτικές πρέπει να σχεδιάζονται όχι για να ενισχύουν την ε, μεροληψία αυτή, αλλά για να τη διορθώνουν. Αυτό το bias. Δυστυχώς, με τους ίδιους πόρους αυτό δεν ισχύει. Η συνθήκη πώς χρηματοδοτείται η Ευρωπαϊκή Ένωση εθνικού προπολογισμού ενισχύει αυτή τη μεροληψία και σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν βοηθά στη διόρθωσή τη. Δημιουργεί δηλαδή ένα zero-sum game αν θέλετε. Έχουμε το σύστημα των ιδιών πόρων στην Ένωση το οποίο γίνεται αντιληπτό ως ε, ένα σύστημα που έχει κάποιους κερδισμένους και κάποιους χαμένους. Ότι δεν υπάρχει δηλαδή μια σωστή ανακατανομή πλούτου αλλά ότι μεταφέρεται πλούτος κάποιων κρατών σε κάποια άλλα και δημιουργείται τελικά αυτό που θα μπορούσαμε να ορίσουμε ως δημοκρατική γνωστική στρέβλωση για όλους αυτούς. Το Zero Sum Game που είπα, το ότι η Ένωση θεωρεί ότι ουσιαστικά δεν ε, ανακατανέμει τον πλούτο που δημιουργείται στις ε, αγορές, αλλά από τη μία χώρα στην άλλη. Τι γίνεται και τι θα μπορούσε να γίνει. Θα μπορούσε μια λύση να είναι η διασύνδεση του συστήματος ιδίων πόρων σε δραστηριότητες που θα μπορούσαν να ασχοληθούν με δύο πτυχές. Το πρώτο, οικονομική δραστηριότητα, που είναι δυνατή μέσω της ε, εσωτερικής αγοράς Όσο περισσότερο οι χρηματοπιστωτικοί πόροι της Ένωσης ε, συνδέονται με τον πλούτο που οι πολίτες σχετίζουν με οικονομικές δραστηριότητες που καθιστά εφικτές η εσωτερική αγορά, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η νομιμοποίηση αυτής της χρηματοδότησης. Δεύτερη πτυχή. Εάν το συσχετίσουμε με τον πλούτο που δεν μπορεί να φορολογήσουν αποτελεσματικά τα κράτη-μέλη, με άλλα λόγια, ε, τα οικονομικά της Ένωσης σχετίζονται με την διόρθωση της φορολογικής ανισότητας και αδικίας με την ε, νέα, ε, με την ε, νέα εξισορρόπηση και μεγαλύτερη φορολογική δικαιοσύνη είναι θετικό και μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει και το αφήγημα ότι ελαφρύνει το φορολογικό βάρος γιατί υπάρχει αυτή η διόρθωση της φορολογικής αδικίας που βλέπουμε σε εθνικό επίπεδο ε, σε ευρωπαϊκό. Αυτό το έλεγε και ο κύριος Φερνάντες. Δηλαδή φαίνεται ότι έτσι αναδιανέμεται ο πλούτος ε, και αποκαθίσταται η φορολογική δικαιοσύνη. Αυτό δίνει μεγαλύτερη νομιμοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα βρει και έτσι και μεγαλύτερη υποστήριξη ε, η Ένωση από τους πολίτες. Το δεύτερο που κάναμε στην έρευνα ήταν ακριβώς να δοκιμάσουμε αυτή την υπόθεση. Αν αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτείται η Ένωση, αλλάζει η αντίληψη των πολιτών για την Ευρωπαϊκή Ένωση και υποστήριξε τις προσοικονομικές πολιτικές της. Θα σας πω ποιες είναι οι ε, εντυπώσεις μας και ποια είναι τα αποτέλεσματα στα οποία καταλήξαμε. Πρώτα απ' όλα, ένα ερώτημα που θέτουμε είναι επειδή έγινε και από τη Γιούγκοβ μεγάλη ε, εκπροσώπηση, ε, βέβαια εδώ εκπροσωπείται και ένα κράτος που δεν θα είναι σύντομα, αλλά ε, το ερώτημα ήταν λοιπόν το πρώτο, αν θεωρείτε ότι θα πρέπει να δίδονται περισσότεροι πόροι στην Ένωση και λιγότεροι στα κρατημέλη ή αντιστρόφως ότι θα πρέπει να δίνονται περισσότεροι πόροι στα κράτη-μέλη και λιγότεροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπετε από τις απαντήσεις ότι υπάρχουν και πολλοί που δεν είναι βέβαιοι. Δεν ξέρουν τι να απαντήσουν, αλλά βλέπουμε στο Νότο, όπου οι περισσότεροι θέλουν να, δίνονται περισσότεροι πόροι στην Ένωση και λιγότεροι στα κράτη-μέλη και στα βόρεια κράτη, στα βορειότερα κράτη-μέλη της Ένωσης, σε σχέση και με τη μεροληψία που σας περιέγραψα, αυτό το bias, οι πολίτες περισσότερο θα ήθελαν ε, οι πόροι να πηγαίνουν στα κρατημέλη και λιγότεροι πόροι ε, στην Ένωση, με εξαίρεση στη Γερμανία όπου εκεί ο κόσμος πιστεύει ότι τα κράτη-μέλη ε, θα έπρεπε να έχουν παίρνουν λιγότερους πόρους και η Ένωση περισσότερο. Υπάρχει όμως αυτή η διαίρεση βορρανότου. Και αυτή η διαίρεση εξαφανίζεται σχεδόν, θα έλεγα, και υπάρχει υποστήριξη χρηματοδότησης προς την Ένωση που αυξάνεται πολύ, αν μπει τελείως διαφορετικά, αν τεθεί τελείως διαφορετικά το ερώτημα. Δηλαδή, αν ρωτήσουμε τους πολίτες αν θα στήριζαν ένα νέο φόρο για τον άνθρακα, για παράδειγμα, εκεί βλέπουμε σχεδόν ε, συνολική υποστήριξη από όλα τα κρατη Το βλέπετε. Αν θα υποστήριζαν το, τη φορολόγηση μεγάλων, ε, παραδείγματος χάρη, Ιντερνετικών πάλι το ίδιο. Και το ίδιο αν και όχι σε τόσο ε, ολικό. Είναι για τους φόρους ε, των ε, εταιριών, Να ξέρεις κάποιες σκανδιναβικές χώρες που υπάρχουν εδώ περισσότερες αμφιβολίες για έναν εταιρικό φόρο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όλα αυτά όμως τι δείχνουν. Δείχνουν ότι τελικά αυτή η υπόθεση Δηλαδή ότι αν αλλάξει ο τρόπο χρηματοδότηση Ένωση, αν έχουμε τότε από εθνικού προπολογισμού να χρηματοδοτείται από του ιδίου πόρου, τότε αν ισχύει αυτό η υπόθεση, αυξάνεται και η υποστήριξη για τη χρηματοδότηση στην Ενωσιακή, αλλά και ε, η στήριξη των πολιτικών τη Ένωση και η νομιμοποίηση τη Ένωση. Δεν θέλω να υπερβώ πάρα πολύ το χρόνο, απλά σα το λίγη υπομονή ακόμη, ε, για λίγα λεπτά ακόμη. Ένα άλλο θέμα που είδαμε κατά πόσον οι ίδιοι πόροι μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτική αντί τη φορολογική εναρμόνιση. Και σχετίζεται και με τα προηγούμενα ε, στοιχεία τα οποία σα έδειξα και τι προηγούμενε ερωτήσει που θέσαμε. Νομίζω ότι θα ήταν δυνατόν και είναι κάτι που θα πρέπει να εξεταστεί ω ενδεχόμενο. Αντί δηλαδή να προσπαθούμε κάτι που είναι δύσκολο, το ξέρετε όλοι, δηλαδή την εναρμόνιση του εταιρικού φόρου για παράδειγμα, των εταιρικών φόρων να επιτρέψουν το φορολογικό ανταγωνισμό, όμως να ε, προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε έναν εταιρικό φόρο για κάποιο επίπεδο εναρμόνισης. Ουσιαστικά αυτό που προτείνουμε είναι να επιτραπεί ο φορολογικός ανταγωνισμός, αλλά να ορίσουμε ότι δεν μπορεί κανείς να πάει κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο, επίπεδο, κατώτατο φορολογικού ανταγωνισμού. Γι' αυτό χρειάζεται μια κοινή ε, βάση ε, φορολόγησης εταιριών, η οποία μπορεί να επιτρέψει και κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι ενδιαφέρον να δοκιμάσουμε και να εξετάσουμε ως ενδεχόμενο σε αυτή την περίπτωση. Υπάρχει αυτό το επίπεδο που θα λέω ότι θα πρέπει να ισχύει παντού για να μην υπάρχει στρέβλωση ανταγωνισμού. Αν έχουμε αυτή την κοινωνιοποιημένη φορολογική βάση, θα μπορούσαμε να ε, δούμε τι διασυνοριακές ε, δραστηριότητες υπάρχουν και τι εθνικές δραστηριότητες υπάρχουν. Αν εφαρμοστεί σε όλες τις δραστηριότητες, αυτό το φορολογικά έσοδα που θα προκύπτουν από τα εθνικά ε, έσοδα διαχωρίζεται από τα έσοδα τα οποία είναι εντός εγωικών ευρωπαϊκά και μπορούν να χρηματοδοτήσουν τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Αυτά είχα να πω ευχαριστώ και συγγνώμη που ξεπέρασα το χρόνο κατά δύο λεπτά. Thank you, uh, Professor Maduro. Uh, Ευχαριστούμε κύριε Μαδούρο, ευχαριστώ και τον καθηγητή Άντορ για την ε, προηγούμενη παρουσίαση. Τώρα να περάσουμε στις ε, ερωτήσεις και στα σχόλια των ε, συναδέλφων. Όμως ε, θα πρότεινα πρώτα να ακούσουμε τις ερωτήσεις και μετά να δώσουμε το λόγο στους προσκεκλημένους προκειμένου να απαντήσουν ε, με έναν ε, συνοπτικό τρόπο. Ας ακούσουμε τους σκιόδης καταρχήν, κυρία Γκουελμίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγγνώμη γιατί έφτασα καθυστερημένη. Δεν μπόρεσα λοιπόν να ακούσω την πρώτη παρουσίαση. Βέβαια, άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά τη δεύτερη. Και σκεφτόμουν πόσο ικανοποιητικά μας παρουσίασε τα επιχειρήματα του κ. Μαδούρο. Εμείς έχουμε ένα position paper ως ομάδα των σοσιαλιστών, ε, ελπίζοντας ότι η επέκταση των ιδίων ε, πόρων ε, θα αποτελέσει ένα πραγματικό στόχο αυτής ε, της θητείας και θα εφαρμοστεί πλήρως σε σύνδεση και με τις διαπραγματεύσεις της ευρύτερες για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Όπως μας παρουσιάσατε κι εσείς βάσει κάποιων στοιχείων και εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να προωθήσουμε αυτή την αλλαγή παραδείγματος και να αυξήσουμε την νομιμότητα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων εισάγοντας ε, ένα γνήσιο σύστημα ιδίων πόρων το οποίο θα μας επιτρέψει να μειώσουμε τις ε, εισφορές των μονομένων κρατών μελών βάσει καθάριση του εθνικού εισοδήματος. Πιστεύω λοιπόν ότι τα επόμενα έτη θα πρέπει να εφαρμόσουμε αυτές τις αλλαγές, αυτή την αλλαγή παραδείγματος, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι τις τελευταίες δεκαετίες εμείς ε, ως ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δράσαμε ε, ακριβώς ε, με τον αντίθετο τρόπο όπως δηλώνει η συνθήκη. Γιατί η συνθήκη σαφέστατα δηλώνει ότι οι ευρωπαϊκές δημόσιες πολιτικές και οι στόχοι πολιτικής θα πρέπει να χρηματοδοτούνται κυρίως από ιδίους πόρους και όχι από εισφορές ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος. Αν δείτε όμως τα δεδομένα, θα δείτε ότι ακριβώς το αντίθετο συνέβη τα τελευταία 30 χρόνια θα έλεγα. Έτσι λοιπόν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να ανατρέψουμε αυτή τη λογική και να έχουμε ένα νέο γνήσιο σύστημα ιδίων πόρων. Εγώ θα ήμουν υπέρ ε, του να έχουμε τη σύνδεση μεταξύ ιδίων πόρων και της εσωτερικής αγοράς και ακριβώς εσείς μας δείξατε ότι οι πολίτες ε, πραγματικά έχουν ε, ευαισθησία απέναντι και συνειδητοποιούν τη λειτουργία της ενίας αγοράς και συνειδητοποιούν ότι τους φέρνει ευημερία η εσωτερική αγορά. Επίσης συνειδητοποιούν και τι συμβαίνει με την κλιματική αλλαγή. Επομένως, ε, προβληματιζόμαστε για ένα νέο, καλά, συγγνώμη, σκεφτόμαστε πια ενός ε, νέου καλαθιού για τους ε, ιδίους πόρους. Πραγματικά εξεπλάγει από τα δεδομένα σχετικά με το φόρο επί του άνθρακα. Μας είπατε ότι οι πολίτες θα συμφωνούσαν με την εισαγωγή ενός τέτοιου φόρου όπως συχνά συμβαίνει, ξέρετε, οι πολίτες είναι πιο προοδευτικοί από ότι εμείς που χαράσουμε την πολιτική, από εμά τους πολιτικούς. Επομένως, θα πρέπει να είμαστε πολύ φιλόδοξοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πολύ θαραλέοι για να εισάγουμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Επίσης, θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα είναι και τόσο ενθουσιώδη ε, στο να εισάγει μια ευρία γκάμα ιδίων πόρων, ε, κυρίως επικεντρώνει τη συζήτηση στο φόρο στα πλαστικά και στο σύστημα εμπορία εκπομπών. Αλλά εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο θεραλέοι. Και έχω και μια ερώτηση για τον καθηγητή Μαδούρο. Θέλω να σας ρωτήσω, τι πιστεύετε για την εισφορά της ενιαίας αγοράς γιατί υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις για το θέμα αυτό. Αν έχετε κάποια άποψη λοιπόν θα σας ευχαριστούσα και σας ευχαριστώ και πολύ για την παρουσίασή σας. Ο κύριος Παπαδημούλης. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους εισηγητές και να συμφωνήσω με την εισαγωγική παρατήρηση του κυρίου Μαδούρο ότι έχουμε αρχίσει να το συζητούμε αυτό το θέμα χρόνια και είναι καιρός πια να προσανατολιστούμε σε αποφάσεις. Και επειδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομίζω ότι είναι στην πρωτοπορία αυτής της συζήτησης πιέζοντας την Κομισιόν και το Συμβούλιο να ανοίξει ουσιαστικά το θέμα των ιδίων πόρων, θα ήθελα να πω δύο πράγματα για να είμαι σύντομος. Το πρώτο, συμφωνώ με την συνάδελφο που μόλις μίλησε, ε, η οποία σημειώνει ότι είναι και θεσμική υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναπτύξει την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των ιδίων πόρων. Αυτή η πολιτική ιστορική εκκρεμότητα είναι σε αντίθεση με αυτό που προβλέπουν οι συνθήκες. Αυτό που γίνεται τώρα είναι αντικανονικό. Να είναι το μεγάλο κομμάτι της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη συμβολή των κρατών μελών και όχι από ίδιους πόρους. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Ε, είχε φτιαχτεί στο παρελθόν μια επιτροπή σοφών. Ονομάστηκε Επιτροπή Μόντι. Αυτή η επιτροπή κατέθεσε ορισμένες προτάσεις για την ανάπτυξη και την ενίσχυση ορισμένων ιδίων πόρων. Θα ήθελα να ρωτήσω και τους δύο εισηγητές πώς αξιολογούν αυτές τις προτάσεις. Είναι καλές προτάσεις, πρέπει να τις ενισχύσουμε, πρέπει να τις βάλουμε σε εφαρμογή. Και το δεύτερο που θα ήθελα να το θέσω υπόψη της δικής μας Επιτροπής, ε, κύριε Όβερβελτ, και υπόψη όλων των μελών της ε, Επιτροπής Budget του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι μετά από αυτό το hearing τι, ποια είναι η δική μας η συνέχεια, το follow-up μετά από αυτό το hearing. Η, η πρότασή μου είναι να σκεφτούμε πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να ανεβάσει πιο ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων το θέμα των ιδίων πόρων με δικές μας προτάσεις που να αξιοποιούν και τη συμβολή των ειδικών, καθώς είναι ολοφάνερο ότι αυτό συνδέεται και με την συζήτηση και τη διαπραγμάτευση για το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Γιατί αν ενισχυθούν οι ίδιοι με προτάσεις που μπορούν ε, να συγκεντρώσουν πλειοψηφίες, τότε θα μειωθεί η πολιτική διαμάχη που συχνά οδηγεί σε αδιέξοδα ανάμεσα στους net contributors και τους net receivers η οποία διαμάχη ανάμεσα στα κράτη-μέλη καθαρούς εισφορείς και καθαρούς λήπτες οδηγεί στο τέλμα. Οδηγεί σε αυτό που ζούμε ήδη εδώ και καιρό να έχουμε ένα συμβούλιο το οποίο αποτελεί φρένο και εμπόδιο στο να καταλήξουμε σε ένα φιλόδοξο πολιετή προϋπολογισμό όπως τον θέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα η πρότασή μου είναι να δώσουμε μια συνέχεια σε αυτό το hearing και να πάρουμε εμείς πρωτοβουλία ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να καταθέσουμε προτάσεις στο θέμα των ιδίων πόρων. Ευχαριστώ. Thank you. Uh, Mr. Ευχαριστούμε, κύριε Φερνάντες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, δύο ομιλητές ε, και κυρίως ε, ο κύριος ε, Μαδούρο μας ενθάρρυνε και μας ενέπνευσε. Η ερώτησή μου είναι, εντάξει έχουμε πείσει τους πολίτες, τα κράτη-μέλη πώς θα τα πείσουμε. Γιατί βλέπουμε μεγάλο δισταγμό από τα κράτη-μέλη, ακόμη και αν γνωρίζουν ότι οι πολίτες ε, είναι θετική έτσι ώστε οι φόροι και για να έχουμε φορολόγηση και να καταπολεμήσουμε την φοροδιαφυγή. Οι πολίτες ε, είναι θετικοί. Ακόμη και για το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών λέει οι πολίτες ότι είναι καλή ιδέα. Για τον άνθρακα το ίδιο, για τη φορολόγηση των ψηφικών εταιριών είναι καλή ιδέα. Και την υπερασπίζουν ευρέως. Αυτό δεν μπορούσε ε, μάλιστα και να τους ανακουφίσει. Και εγώ θεωρώ ότι είναι ένα καλό μήνυμα και κατά ε, των ε, λαϊκιστών γιατί οι λαϊκιστές θα πούνε θέλουν να αυξήσουν τους φόρους όμως είναι λάθος αυτό, είναι ψέμα και θα τους διαψεύσουμε πώς μπορούμε να πείσουμε όμως τα κράτη-μέλη και τα εθνικά κοινοβούλια τελικά θα πρέπει να συμφωνήσουν για το τι μπορούμε να κάνουμε παραπάνω. Πώς θα τους πείσουμε. Εγώ έχω παντότε την εντύπωση και ήδη το έχω πει δημοσίως αυτό κάποια φορά, ότι όταν καλέσω κάποιον σε δείπνο και ε, έχω το δικαίωμα να διαλέξει το εστιατόριο και το μενού. Παραδείγματο χάρη η Γαλλία και η Γερμανία είναι υπεύθυνε για το 38% του προπολογισμού. Υπάρχουν κράτη-μέλη που θέλουν να διατηρήσουν ε, με τη βία αυτό το πρόγραμμα. Και ουσιαστικά μειώνοντας ε, τα έσοδα που έρχονται από τους εθνικούς προϋπολογισμούς ε, σε κάποια κράτη-μέλη μπορεί να θεωρείται ότι θα έχουν πιο δύναμη θέση στις διαπραγματεύσεις. Όμως θα πρέπει να τα πείσουμε αυτά τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να καταθέσουμε εμεί και κάποιε προτάσει από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να προχωρήσουμε σε μια πρόταση που να πείσει το Συμβούλιο. Ευχαριστώ, κύριε Μάρκες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ καταρχήν ε, θέλω να ευχαριστήσω τους δύο μιλητές ε, για τις παρουσιάσεις τους. Εμείς ε, που διαπραγματευόμαστε το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και τους ίδιους πόρους είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και ακριβώς θα ξεκινήσω με το σημείο αυτό. Δηλαδή, βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο να συζητάμε την κατάσταση των ιδίων πόρων. Αυτό πιστεύω ότι εμείς, ε, το Κοινοβούλιο, θα πρέπει να θέσουμε στη συζήτηση είναι το εξής. Τι σημαίνει για μας να λέμε ότι εμείς ε, θα χαιρετήσουμε τη συνένεση επί του πολιτισμού δημοσιονομικού πλαισίου αν έχουμε και συμφωνία για τους ίδιους πόρους. Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε προώθηση της ε, συζήτησης για τους ίδιους πόρους εγκαίρως ε, πριν να εγκρίνουμε το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και η έννοια της συγκατάθεσης είναι πολύ σημαντική. Σχετίζεται με τη συζήτηση που είχαμε εδώ. Δηλαδή, προφανώς, ε, έχουμε ε, ήδη ε, το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα, το οποίο ουσιαστικά έχει ένα μη ισορροπημένο βάρος σε σχέση με την χρηματοδότηση μέσω ιδιών Και αυτή την τάση εμείς θέλουμε να αλλάξουμε και γι' αυτό πιστεύω ότι συμβιβασμός απαραίτητα θα πρέπει να βρεθεί εδώ, να έχουμε ένα πολιτικό συμβιβασμό, δηλαδή ότι θα αυξηθεί η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των ιδίων πόρων. Ίσως ε, θα ε, μπορούσε να είναι λανθασμένη ε, η ερμηνεία, όμως δεν θέλουμε να αλλάξουμε την ισορροπία. Πρέπει να αυξηθεί η χρηματοδότηση. Και εφόσον εμείς συμφωνούμε με τις πολιτικές αρχές, ακόμη και το Συμβούλιο συμφωνεί με τις πολιτικές προτεραιότητες του Κοινοβουλίου, κατόπιν όμως βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη στάση. Τώρα, το δεύτερο σχόλιο έχει να κάνει με κάτι που έθιξε και ο κύριος Φερνάντες. Δηλαδή, ότι αυτοί οι νέοι ήδη πόροι θα μπορούσαν να σημαίνουν μεγαλύτερη φορολογική δικαιοσύνη, γιατί ταυτόχρονα θα συνεισφέρουν στην καταπολέμηση της φοροαπηγής και της φοροδιαφυγής. Επομένως, είναι σημαντικό να δώσουμε αυτή την εξήγηση ότι εδώ δεν θέλουμε να επιβάλλουμε πρόσθετους φόρους στους πολίτες είναι ένα ε, θέμα πολιτικής εκπροσώπησης που έθεσε ο κύριος Μαδούρο. Δηλαδή, σε σχέση με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η εκπροσώπηση των πολιτών γίνεται σε δύο επίπεδα. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε άμεση εκπροσώπηση και στο Συμβούλιο έχουμε έμεση εκπροσώπηση μέσω των κυβερνήσεων. Επομένως, εμείς στην πολιτική εκπροσώπηση έχουμε την εκπροσώπηση και των κρατών και των πολιτών και επομένως αυτή η εκπροσώπηση επίσης θα πρέπει να μεταφερθεί και στην συμμετοχή με οικονομικούς όρους. Και εξηγώ τι σημαίνει αυτό, ότι θα πρέπει να αυξηθεί η ατομική εισφορά των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτο σημείο, μια ανησυχία θέλω να εκφράσω εδώ. Στη συζήτηση αυτή, κατά τη δική μου άποψη, εμείς θα πρέπει να αποφύγουμε ε, και θα χρησιμοποιήσω την αγγλική έκφραση taxes oriented. Εμείς δηλαδή ε, δεν συζητάμε τους ίδιους πόρους και τον κάθε πόρο που θα είναι προγραμματισμένος, προσανατολισμένος σε μια πολιτική. Δεν μπορούμε να έχουμε δύο σπόρους που να συνδέονται το χάρη με τον Green Deal που θα χρηματοδοτήσουν τον Green Deal. Εγώ νομίζω ότι το θέμα των ιδίων πόρων θα πρέπει να ειδωθεί από μια πτυχή, από μια σκοπιά ενότητας και ολότητας, καθολικότητα του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, και σε αυτά τα θέματα θα ήθελα να ακούσω τα σχόλιά σα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Madame Holmeier. Κυρία Χολμάιερ. Ε, Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ Πρόεδρε, αυτό το οποίο έτσι με ε, εντυπωσιάζει σε αυτή τη συζήτηση είναι ότι είμαστε υπέρ ε, το να έχουμε περισσότερα έσοδα, αλλά υπάρχει αυτή η άποψη τα κράτη-μέλη είναι κακά, κανείς δεν θέλει να πληρώσει, δεν μπορεί να συμφωνήσουν μεταξύ τους. Τελικά είναι μια στρατηγική αυτή, γιατί όλοι ξέρουμε ότι ο άλλος είναι ο κακός, ο άλλος τα κάνει άσχημα και τελικά Πού καταλήγουμε πουθενά με αυτή τη συζήτηση σε ό,τι δεν αφορά ε, τη φορολογία. Ξέρουμε ότι απαιτείται ε, ομοφωνία ε, και για το ΠΔΠ και για το σύστημα ιδιοπόρων και επομένως μπορούμε να τα σκεφτούμε όλα αυτά, αλλά σίγουρα και το είπε και σωστά ο συνάδελφος Μερνάντες ε, πρέπει κάπως να προσετεριστούμε τα κράτη-μέλη, να τα φέρουμε πιο κοντά στα νερά μας, να καταλάβουν ε, τι ε, πρέπει να γίνει. Σίγουρα υπάρχουν έσοδα που ε, γυρίζουν πίσω στα κράτη-μέλη και όχι σε εμά. Ε, αν θέλουμε τα δικαιώματα εμπορίας εκπομπών, αυτό το σύστημα να το διευρύνουμε, θα πρέπει να ασχοληθούμε πολύ περισσότερο με το θέμα της πράσινη Συμφωνίας και πρέπει να τονίσουμε και την ανάγκη να υπάρξει επέκταση του συστήματο των ιδιών πόρων. Το δεύτερο, μου άρεσε και εμένα πολύ ε, η παρουσίαση που άκουσα. σίγουρα, όταν ένας πολίτη ερωτηθεί ε, για ένα φόρο που αφορά έσω τους άλλους, ε, δεν είναι κατά, φυσικά και είναι υπέρ. Αν χάνει έσοδα, ε, θα είναι κατά. Υπάρχει δηλαδή ουσιαστικά ένα ερώτημα το οποίο γυρίζει πίσω συνεχώς. Το θέμα είναι η λογική χρηματοδότηση. Πώς μπορεί να είναι λογικές οι προτάσεις σε ό,τι αφορά την απάτη, ε, σε ό,τι αφορά ε, δασμούς ή το ΦΠΑ, ε, από αυτά, από την απάτη, χάνουμε πολύ περισσότερα. Αν αυτό ε, το καταλάβουν οι πολίτες, νομίζω ότι θα αλλάξει πάρα πολύ και η όλη συζήτηση 3,5 δις ήταν τα διαφυγόντα κέρδη μόνο από μία υπόθεση ε, και φανταστείτε τι γίνεται συνολικά εάν και οι τελωνιακές αρχές δραστηριοποιηθούν ακόμη περισσότερο ε, και αν ελέγχονται περισσότερα προϊόντα ε, τα οποία εκτελονίζονται. Νομίζω ότι και πολλά προβλήματα μπορούμε να αποφύγουμε. Σίγουρα έχουμε δηλαδή και εδώ ανάγκη να ενισχύσουμε το έργο μας ε, για τους ιδίους πόρους, ε, φυσικά και θα πρέπει να το συζητήσουμε. Αλλά πρέπει να δούμε με ποια εργαλεία μπορούμε να έχουμε επιτυχία. Και όχι να λέμε απλά αγωνιστήκαμε, παλέψαμε, αλλά δεν πετύχαμε τίποτα. Αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα. Πρέπει να επιδιώξουμε λύσεις που είναι φυκτές και στα κράτη-μέλη που δεν θα αρχίσει ο καθαρός συνεισφέρον να, τα ρίχνει στον καθαρό δικαιούχο και τούμπαλιν ε, και να υπάρχει αντιπαράθεση μεταξύ αυτών των δύο κατηγοριών. Και από κοινού ε, θα πρέπει να το παλέψουν, γιατί ξέρετε ότι και στις χώρες μας δεν συμφωνούμε όλοι για το 1,3%. Υπάρχουν και κάποιοι που είναι υπέρ του 1,1 ή του 1,0 κάτι. Επομένως, ας τα δούμε όλα αυτά ε, και να δούμε τι γίνεται και ε, στα Εθνικά Κοινοβούλια. Ε, θα έπρεπε όλοι να συζητήσουμε με τους συναδέλφους μας και σε εθνικό επίπεδο. Πρέπει να δούμε τι γίνεται, ποιες είναι οι απόψεις για τα έσοδα, για τις δαπάρες. Εμείς δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τους, τις εθνικές κυβερνήσεις και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Οι συνάδελφοι στις χώρες μπορούν. Κυρία Κέλλερ έχει τώρα το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παίρνω και εγώ το λόγο μετά τα όσα είπαν οι προλαλήσαντες και συμφωνώ μαζί τους. Θέλουμε να έχουμε γνήσιους ιδίους πόρους, θα πρέπει να έχουμε τα απαραίτητα μέσα για να το πετύχουμε αυτό. Παίρνοντα λοιπόν αυτή τη στιγμή το λόγο, θα ήθελα να μιλήσω λίγο περισσότερο για αυτό το μηχανισμό συμπερίληψη του άνθρακα στα σύνορα. Θεωρώ ότι έχει δύο θετικά ένα τέτοιο μηχανισμό. Από τη μία πλευρά, αποτρέπει την διαρροή άνθρακα, το λεγόμενο carbon leakage, ουσιαστικά ζητώντας την καταβολή του περιβαλλοντικού κόστους σε σχέση με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ πέρα έχουμε από τη μία την τιμή του ETS, δηλαδή την τιμή που πρέπει να πληρώσουν οι εταιρείες όσον αφορά τα δικαιώματα εμπορίας εκπομπών και από την άλλη όμως πρέπει να καταβάλουν και τη διαφορά της τιμής άνθρακα από τη μία χώρα στην άλλη. Ο μηχανισμό λοιπόν αυτό που δεν θέλω να αποκαλέσω φορολογικό μηχανισμό μπορεί να είναι ιδιαίτερα θετικό και για το περιβάλλον αλλά και για την αύξηση των εσόδων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι θα πρέπει πολύ γρήγορα να εξετάσουμε τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιήσουμε για την εφαρμογή του κανονισμού αυτού. Γιατί έχει να κάνει και με τα πρωτογενή προϊόντα αλλά και με τα μεταποιημένα προϊόντα τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν σε αυτό το μηχανισμό. Και χαίρομαι γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε πολλά θετικά στατιστικά δεδομένα μας λένε ότι πάρα πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες θέλουν τους φόρους αυτούς. Δυστυχώς όμως κάθε φορά που μιλάμε εμπράκτος για τα ζητήματα αυτά υπάρχουν πολλές ενός καταναλωτών που αρχίζουν και στρέφονται κατά των ιδεών αυτών και επηρεάζουν εν γέννη και την κοινή γνώμη τότε. Γιατί στη τελευταία ανάλυση πάντα ο καταναλωτή καταβάλει το, το τίμη μα, μην γελιόμαστε. Θα μπορούσατε λοιπόν και απευθύνομαι αυτή τη στιγμή στα μέλη του πάνελ Ποια διαδικασία θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε προκειμένου να προχωρήσουμε λίγο περισσότερο προς την υλοποίηση αυτού του μηχανισμού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και εσείς κύριε καθηγητά θα μπορούσατε να μας μιλήσετε λίγο περισσότερο για την ε, θεωρητική αλλά και την εφαρμοσμένη πτυχή των συστημάτων αυτών φορολογίας και πώς αυτή γίνεται αντιληπτή ή αποδεκτή από τους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστούμε κύριε Καρθιαμπάλη, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και τους ομιλητές μας για τις ιδέες τους, για τις προτάσεις τους. Έλεγε ο καθηγητής Μαδούρο ότι όταν γινόταν λόγος πριν από ε, κάποια χρόνια για του ίδιου πόρου. Αυτό που μίλαγε για αυτό το θέμα θεωρεί το λίγο πολύ τρελό και έχει αλλάξει βέβαια η κατάσταση τώρα. Φυσικά και είμαστε υπέρ των ίδιων πόρων, βλέπουμε τα ωφέλη ε, που έχει το να υπάρχουν πόροι που θα χρηματοδοτούν τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Το θεωρούμε πλέον προφανέ. Αλλά το Συμβούλιο δεν έχει αλλάξει παρόλα αυτά. Και συμφωνώ με τους συναδέλφους που ρώτησαν τι θα κάνουμε για να αλλάξει άποψη το Συμβουλίο. Γιατί όταν μιλάμε ε, με τους πρωθυπουργού ή τους προέδρους των κυβερνήσεων μας λένε πολλές φορές εγώ είμαι υπέρ αλλά δεν θα το δεχτούν οι πολίτες. Άρα οι στατιστικές και οι μελέτες ε, ε, δεν φαίνεται ότι δείχνουν αυτό, δείχνουν το αντίθετο κιόλα από αυτό που ισχυρίζονται οι πολιτικοί. Περάσαμε μια οικονομική κρίση που οδήγησε σε αύξηση του φοροεισοδήματο, αύξηση του ΦΠΑ και δημιούργησε μεγάλη δυσαρέσκεια όλο αυτό βέβαια στου πολίτε. Αυτό μπόρεσαν να το κάνουν οι εθνικέ κυβερνήσει. Και τώρα δεν μπορούμε να επιβάλλουμε του φόρου στου ρηπαίνοντε στι επιχειρήσει που προβαίνουν σε απάτη. έναν κατώτατο εταιρικό φόρο, επιτρέποντας βέβαια τον ανταγωνισμό. Δεν μπορούμε να τον επιβάλλουμε. Άρα τι κάνουμε. Καταλήγουμε στο, στο συμπέρασμα ότι γίνεται μεν κάποιος λόγος στο Συμβούλιο, αλλά δεν προχωρά. Δεν μπορώ να συμφωνήσουν. Ούτε για τις εκπτώσεις, ε, για την κατάργησή τους. Ε, εδώ λέγαμε για προσθήκη ε, φόρων ε, και νέες εισφορές, ε, αλλά όχι απλά αυτό δεν σκέφτονται. Εδώ δεν θέλουν καν να περιορίσουν τις εκπτώσεις και επιστροφές προς πλούσιες χώρες κιόλα. Το θέμα είναι να προχωρήσουμε, αλλά για να προχωρήσουμε πρέπει να πείσουμε τα κράτη να εγκρίνουν ε, πόρους. Υπάρχουν κάποια κράτη επίσης που είναι υπέρ κάποιων νέων πόρων και κάποιων άλλων κατά και τελικά δεν προχωράμε. Εμείς αυτό πρέπει να κάνουμε είναι όλοι να δεχθούν ε, κάποιους ε, φόρους. Κάποιοι είναι πιο ευεργετικοί, κάποιοι λιγότερο. Ε, μπορεί να επηρεάσουν περισσότερο τα ε, έσοδα τα φορολογικά που εισπράττονται. Έχω δύο διευκρινήσεις να ζητήσω ε, πάω περισσότερα πράγματα να ακούσω. Ε, καταρχάς για τους όρους, τις αιρεσιμότητες που μίλησε ο κύριος Άντορ, τα conditionalities αν υπάρχει χρόνος ε, να συζητήσουμε για αυτό το θέμα λίγο πιο διεξοδικά, με συγκεκριμένα παραδείγματα, κύριε Άντορ. Και στον κύριο Μαδούρο το ερώτημα είναι πάνω στο τελευταίο, που πάλι δεν μπορέσετε να αναπτύξετε κι εσείς γιατί δεν είχατε πολύ χρόνο. Αυτό τον εταιρικό φόρο, αυτή την κοινή φορολογική ενωπημένη βάση, πώς θα λειτουργούσε. Υπάρχει κάποια μελέτη ως προς το πόσα θα μπορούσαν να σπραχθούν με αυτό το μέτρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κίρτσος έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ε, νομίζω ότι το βασικό μας πρόβλημα είναι ότι έχουμε το Brexit, δηλαδή φεύγει το Ηνωμένο Βασίλειο, που σημαίνει ότι πρέπει να αναπληρώσουμε ε, πόρους για, την ευρωπαϊκή, για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, αλλά δυστυχώς μένει μαζί μας η νοοτροπία του Brexit. Θα σας θυμίσω ότι η φράση της Θάτσερ που ξεκίνησε τη διαδικασία πριν δεκαετίες βέβαια του αποχωρισμού, ήταν «I want my money back». Και το ακούμε αυτό συνεχώς σε αυτές τις αίθουσε σε διαφορετικές παραλλαγές. Και θα σας πω το εξής, ότι ε, έχουμε μπροστά μας μεγάλες προκλήσεις, οι οποίες είναι πρακτικά δύνατο να χρηματοδοτηθούν. Εχθές ήμουνα στην Επιτροπή ΣΕΝΤΕ και μιλάγαν, <laughs> μιλάγαμε πώς θα πάμε στο 6G γιατί χάσαμε τη μάχη του, 5G, ε, του τηλεπικοινωνικού δικτύου, από τους Κινέζους. Ναι, αλλά οι Κινέζοι για να κερδίσουν τη μάχη του 5G κάνανε επιδοτήσεις και διευκολύνσεις στις τάξεις των 50 με 60 δισεκατομμυρίων ευρώ. Επομένως, πού είναι η χρηματοδότηση για να πάμε στο 6G έχοντας χάσει το 5G. Ή ακόμα η πράσινη μετάβαση, μια, μια προσεκτική ματιά στα, στα χρήματα που δίνονται είναι εντελώς ανεπαρκή, γιατί ουσιαστικά είναι τα περισσότερα είναι χρήματα ε, του προϋπολογισμού από άλλες δράσεις που θα πάνε στην πράσινη μετάβαση. Ή πάμε στην άμυνα. Στην άμυνα, επειδή ασχολούμαι και με αυτά τα θέματα στην Επιτροπή ΣΕΝΤΕ, ε, τέλος πάντων προωθούμε μια αύξηση ε, για πρώτη φορά αμυντικές δαπάνες στη τάξη των 8 έως 11 δις για την επόμενη επταετία. Γίνεται μια, ένας φοβερός καυγάς πώς θα μειωθούν αυτά τα ποσά τα οποία ακόμα δεν έχουν εγκριθεί. Ε, και βέβαια η Κίνα, που είναι η δεύτερη δύναμη σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει αιτήσει ο προπολογισμό στρατιωτικό τη τάξη των 250 δις δολαρίων. Επομένω ο κόσμο έχει αλλάξει, εμεί έχουμε μείνει στα ίδια και πάμε για μια φοβερή κρίση αξιοπιστία, γιατί οι στόχοι που θέτουμε είναι πρακτικά αδύνατο να χρηματοδοτηθούν με αυτά που συζητάμε. Ε, επειδή προέρχομαι από την Ελλάδα και ορισμένοι θα σκέπτονται ότι τέλος πάντων θέλω, προσπαθώ να αποσπάσω ορισμένα πρόσθετα κονδύλια για να βοηθήσω τη χώρα μου που έχει πρόβλημα αναπτυξιακό, κοινωνικό και διάφορα άλλα, θα σας πω ότι εδώ χρειαζόμαστε μια κοινή προσπάθεια να αυξήσουμε τους ίδιους σπόρους και να δεσμευτούμε ότι θα πάνε σε νέες πολιτικές. Διαφορετικά, οι οικονομίες που, νομίζουμε ότι κάνουμε σήμερα, σε πέντε χρόνια θα είναι τεράστιοι λογαριασμοί, γιατί θα έχουμε πέσει πίσω σε όλους τους τομείς ε, στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Άλλωστε αυτά που συμβαίνουν από τη Συρία μέχρι τη Λιβύη όπου διάφοροι πρωταγωνιστούν επειδή εμείς είμαστε εντελώ απόντες ενώ σαν Ευρωπαϊκή Ένωση μας προειδοποιούν για τους κινδύνους. Άρα θα ήθελα προτάσεις ή μάλλον θα ήθελα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λέει όχι ε, σε αποφάσεις που δεν χρηματοδοτούνται. Ε, είναι ένας κανόνας που ισχύει στα εθνικά κοινοβούλια. Νομίζω μπορούμε να το κάνουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. thank you. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Άντερσεν. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτό το παράθυρο ευκαιρία που ανοίγεται, καθότι βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, πολλοί Ευρωπαίοι πολίτε που αυτή τη στιγμή τίθενται υπέρ τη χρησιμοποίηση περισσότερων ιδίων πόρων για τον κοινοτικό προπολογισμό. Η υποστήριξη υπάρχει και από ορισμένε κυβερνήσει και αυτό είναι θετικό. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει και εμεί να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι, λιγότερο θεωρητικοί. Δεν αρκεί πλέον να λέμε χρειαζόμαστε περισσότερου γνήσιου ή ίδιου πόρου. Πρέπει να λέμε συγκεκριμένα ποιου ίδιου πόρου θέλουμε, πώ θα καταφέρουμε να του καταρτήσουμε. Για παράδειγμα, ο διαστονοριακός φόρος όσον αφορά τον άνθρακα θα μπορούσε να ήταν μια πάρα πολύ καλή πηγή εσόδου για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένας νέος γνήσιος τρόπος χρηματοδότησης του νοσιακού προπολογισμού που μάλιστα δεν προκύπτει μεμονωμένα από ένα κράτος μέλος αλλά προϋποθέτει τη συλλογικότητα, τη συμμετοχή πολλών κρατών μελών και μάλιστα λειτουργεί και υπέρ του περιβάλλοντος. Συζητώντας λοιπόν ένα τέτοιο διασυνωριακό φόρο άνθρακα ακούμε δύο ήδη επιχειρημάτων και θα ήθελα εδώ πέρα τη γνώμη των εμπειρογνωμόνων μας. Πρώτον, υπάρχουν ορισμένοι που μας λένε ότι με ένα τέτοιο φόρο θα έχουμε πρόβλημα με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Ορισμένοι λένε ότι δεν μπορεί κανείς να επιβάλλει ένα τέτοιο φόρο για τον άνθρακα, γιατί θα έρχεται σε αντίθεση με τα όσα ισχύουν για το διεθνέ εμπόριο. Άλλοι πάλι λένε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και ότι ένα τέτοιο φόρο θα μπορούσε να ήταν συμβατό. Ένα δεύτερο επιχείρημα που ακούμε είναι ότι ε, δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή πόσα χρήματα θα καταφέρουμε να αντλήσουμε από ένα τέτοιο φόρο. Εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να επεξεργαστούμε, να διερευνούμε περισσότερο τη δική μα την επίσημη θέση για το φόρο αυτό και προφανώ χρειαζόμαστε τη δική σα τη συμβολή. Η κυρία Αγιέ έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και τους εμπειρογνώμονές μας για τις εξαιρετικές αυτές πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις τους, κάποιες πρώτες δικές μου αντιδράσεις και κάποιες ερωτήσεις εν συνεχεία. Κύριε Άντορ, εσείς αναφερθήκατε στο ζήτημα της χρηματοδότησης του New Green Deal και μας είπατε ότι δεν θα πρέπει να βασιστεί μόνο στον ενωσιακό προπολογισμό η χρηματοδότηση αυτή. Προφανώς συμφωνώ μαζί σας και αν έπρεπε να βασιστεί μόνο στον οσιακό προπολογισμό, τότε το New Green Deal δεν θα ανταποκρινόταν προφανώ στι φιλοδοξίε που έχουμε ήδη εμεί θέσει. Και θα πρέπει να γνωρίσουμε επίση και πώ θα χρηματοδοτεί το στην πράξη μέσω του νοσιακού προπολογισμού του New Green Deal. Όσον αφορά την φορολογική βάση στην οποία αναφέρθηκε η Μόνικα Χολμάιερ, προφανώς δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε περαιτέρω τους Ευρωπαίους πολίτες με ακόμα περισσότερους φόρους. Σε τελευταία ανάλυση, όπως πολύ σωστά είπατε, το τίμημα, τον τελικό φόρο καταβάλει ο Ευρωπαίος πολίτης. Η Ευρωπαϊκή όμως Ένωση και όλοι είμαστε υπέρ, περισσότερο τουλάχιστον υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ πέρα, θα πρέπει να λειτουργεί θετικά, επικοδομητικά, να δημιουργεί ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Με αυτή η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία μέσω των νέων αυτών ιδίων πόρων μπορεί να προκύψει. Και αυτό έχει φανεί και στις δημοσκοπήσεις στις οποίες ανέφερε και ο κύριος Μαδούρο. Οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι δεκτικοί αυτή τη στιγμή, μπορούν να φουγκραστούν τα όσα τους λέμε εμείς. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τη θετική αυτή ευκαιρία που έχουμε και νομίζω ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα νέο καλάθι νέων ιδίων πόρων για τον κοινοτικό προπολογισμό και για τη βιωσιμότητα του προπολογισμού, αλλά και για να αντιμετωπίσουμε τα εμπόδια τα οποία έχουμε μπροστά μα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν κράτη-μέλη που δεν θέλουν ιδίου πόρου, κανένα ίδιο πόρο. Από την άλλη, υπάρχουν όμω κράτη-μέλη που δεν θέλουν, λένε ιδίου πόρου, αλλά από την άλλη μπορεί να πιστούν, μπορούν να προσαρμόσουν την άποψή του, αρκεί να μιλάμε για το κλίμα, μα λένε. Και εσεί, κύριε Μαδούρο, μα είπατε ότι πριν από μερικά χρόνια σας θεωρούσαν ε, αγιατολά πραγματικά σε σχέση με τα όσα λέγατε, ιδιαίτερα ριζοσπαστικό. Αυτή τη στιγμή όμως, από ό,τι φαίνεται, η κοινή γνώμη συμπλέει με τη δική σας την προσέγγιση. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε τη δυναμική αυτή να την, να την χρησιμοποιήσουμε, να την αξιοποιήσουμε. Και ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα χρειαστεί να κάνουμε συμβιβασμούς και εμείς στη συζήτηση που θα κάνουμε το Συμβούλιο, αλλά σε έχουμε τουλάχιστον στο πλευρό μας αυτή τη στιγμή και τους Ευρωπαίους πολίτες. Οι ίδιοι Ευρωπαίοι πολίτες μας λένε ότι θέλουν ιδίους πόρους και μέσω των ιδίων αυτών πόρων μπορούμε να δώσουμε εμείς περαιτέρω πολιτικά κίνητρα. Κύριε Μαδούρο τώρα, θα ήθελα να σας θέσω μία ερώτηση. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά, ακούγοντά σα, όταν μα είπατε ότι το νεύτο καλάθι δύο πόρων θα μπορούσε να αντικαταστήσει το δύσκολο αυτό εγχείρημα τη φορολογική εναρμόνιση. Εγώ νομίζω ότι δεν ασύμβατα αυτά τα δύο. Θα μπορούσαμε να επεξεργαστούμε παράλληλα με διαφορετικά ενδεχομένω χρονοδιαγράμματα. Είπατε επίση ε, όσον αφορά την δραστηριότητα των εταιριών για τις διασυνοριακές οικονομικές δραστηριότητές τους. Αναφέρεστε εδώ πέρα στη διασυνοριακή δραστηριότητα των επιχειρήσεων, έτσι δεν είναι, όχι στα κέρδη τα οποία προκύπτουν στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν βασιζόμαστε μόνο στην εθνική φορολογία, την εταιρική, εκεί πραγματικά δημιουργούμε ανισότητες, καθότι αυτή διαφέρει από τη μια χώρα στην άλλη. Να επανέλθω τώρα στου καθηγητές Άντορ και Μαδούρα για να απαντήσουν και να ακούσουμε και τα προστά σχόλιά τους, κύριο Άντορ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε κάποια σημεία. Πιστεύω ότι με αυτά συνδέθηκε περισσότερο η παρουσίασή μου. Αν δούμε, παραδείγματο χάρη, την έκθεση Μόντι και την αιρεσιμότητα, κυρίως σε ό,τι αφορά την πλευρά των δαπανών και με το πώς θα πείσουμε. Νομίζω ότι είναι μια ερώτηση που θα πρέπει να απαντήσουμε από κοινού με τον κύριο Μαδουρό. Η έκθεση Μόντι μας δίνει ένα ξεκάθαρο κατάλογο συστάσεων και ήδη εγώ βασίστηκα σε μεγάλο βαθμό σε αυτές. Και ανέφερα ότι πρέπει να έχουμε ένα προσανατολισμό προς τα δημόσια αγαθά. Όμως ανέφερα ότι χρειάζεται και κάποια προφύλαξη, κάποια επιφυλακτικότητα, γιατί προκειμένου να είναι νόμιμη η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο προπολογισμό, ε, η εστίαση στα δημόσια αγαθά σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι κάτι πολύ σημαντικό. Απ' την άλλη, να μην υποτιμούμε τις άλλες δύο δημοσιονομικές λειτουργίες, ε, το την αναδιανομητική λειτουργία και τη σταθεροποίηση κυρίως ε, στα πλαίσια μιας νομισματικής ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρώ, θα πρέπει να μπορέσει να κινηθεί και στις ε, τρεις βασικές λειτουργίες αυτές. Όμως, ό,τι αφορά το θέμα της νομιμότητας, ίσως αιτιολογείται να επικεντρωθούμε στα δημόσια αγαθά. Και θα πρέπει να συμφωνήσω με το να υπογραμμίσουμε την κλιματική πολιτική και το Green Deal στο στάδιο αυτό. Πολλοί ομιλητές ρώτησαν πώς θα πείσουμε τους πολίτες, αλλά κυρίως πώς θα πείσουμε τους εθνικούς ηγέτες ε, σε εθνικό επίπεδο. Υπάρχει μια ερώτηση. Αν ε, οι πολίτες ε, βλέπουν ε, τις δαπάνες που συνδέονται με κατηγορίες δαπανών, αν υπάρχει ουσιαστικά ενστερνισμός των κρατικών στόχων. Οι στόχοι που έχουμε στην Ευρώπη δεν αμφισβητούμε και είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι η ευρωπαϊκή δημοσιονομική στόχη δεν θεωρείται ιδιαίτερα ότι υποστηρίζουν τους ίδιους στόχους, αλλά νομίζω ότι βοηθά αν μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι ο ευρωπαϊκός προπολογισμό υποστηρίζει τους εθνικούς στόχους, όπως παραδείγματο χάρη το κράτος πρόνοιας ή άμυνα και ασφάλεια. Επίσης, ε, ε, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δοθεί ότι βοηθά να προωθήσει την τεχνολογική καινοτομία και επίσης να απαντήσει στα θέματα της ε, βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας και ότι οι πόροι βοηθούν στην εφαρμογή των ε, βιομηχανικών πολιτικών. Και αυτό θα βοηθήσει κατά την άποψή μου. Διασυνοριακοί υποδομές τονίζονται επίσης μεταξύ των στόχων να μην ξεχνάμε και το παράδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Η εκστρατεία για το Brexit επικεντρώθηκε σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, μια συνέπεια της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσα θα εξοικονομήσουν αν δεν πληρώνουν στον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Ήταν κεντρικό αυτό το ζήτημα. Γιατί ήταν δυνατό να γίνει αυτό κεντρικό ζήτημα της εκστρατεία, γιατί δεν ήταν ορατό ε, ουσιαστικά ποια ωφέλη λάμβανε το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά λάμβανε πολύ σημαντικά ωφέλη με την πρόσβαση στην ενιαία αγορά και την πρόσβαση σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία δεν είχαν την κατάλληλη προβολή. Έτσι λοιπόν, έχουμε ένα θέμα προβολής, ε, αλλά υπάρχει και ο άμεσος σύνδεσμος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού με τις εθνικές προτεραιότητες. Είναι ένα βασικό σημείο όπου θέλουμε να βασιστούμε και να ενισχύσουμε την υποστήριξη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον περιπλογισμό. Ανέφερα το θέμα της ερεσιμότητας και σε ό,τι αφορά τις δαπάνες συγκεκριμένα, Είπα ότι πιθανότατα θα υπάρχει κάποιος περιορισμός στην ερεσιμότητα, όμως νομίζω ότι ένα σημαντικό τμήμα της πρότασης του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου είναι η σύνδεση με το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Αυτό θεωρείται ένας κύριος διάβλος ε, της ευρωπαϊκής ερεσιμότητας, όμως από αυτή τη σκοπιά ε, θα πείσουμε τους πολίτες, ε, αν δουν και οι πολίτες που οδηγεί το εξάμεινο, ότι δεν είναι απλώς ένα γραφειοκρατικό εγχείρημα που υλοποιεί κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ότι υπάρχουν μακροπρόθεσμοι στόχοι, βιώσιμη ανάπτυξη, στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης ή ακόμη πιο συγκεκριμένα πράγματα στα οποία θέλει ουσιαστικά να μα οδηγήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του εξαμήνου. Διαφορετικά, η νομιμότητα τη αιρεσιμότητα μπορεί να αμφισβητηθεί. Τώρα, πώς θα χρηματοδοτήσουμε την Πράσινη Συμφωνία. Είναι το τελευταίο σημείο που θέλω να απαντήσω. Γιατί είπα ότι ουσιαστικά μικρό ρόλο μπορεί να παίξει ο ευρωπαϊκό προπολογισμό. Μπορεί να παίξει ρόλο αν προσθέσει στου επενδυτικού πόρου ε, στι χώρε και στι περιοχέ συνοχή και να δώσει τα κατάλληλα κίνητρα. Όμω ο ρόλο του τραπεζικού συστήματο είναι θεμελιώδη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την ικανότητα να επηρεάσει τη συμπεριφορά του τραπεζικού συστήματος μέσω των δημόσιων τραπεζών, με τα νέα είδη συνεργασίας μεταξύ των τραπεζών πρόθεσης, promotional banks, κυρίως ε, μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ενοικοδόμησης και Ανάπτυξης. Και εγώ νομίζω ότι αυτός είναι ο πιο εύρωστος διάβλος αν έχουμε το σωστό συντονισμό πολιτικών ε, και ουσιαστικά η Πράσινη Συμφωνία είναι ένα πρόγραμμα επενδύσεων που υποστηρίζεται από πιστώσεις στη σύγχρονη οικονομία και έτσι θα πρέπει ε, ουσιαστικά από τη σκοπιά των δημοσίων πολιτικών να το καθοδηγήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Μαδούρο. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είχαμε πολλές ερωτήσεις, αλλά νομίζω ότι έχουμε δύο μεγάλες ομαδοποιήσεις και έτσι θα προσπαθήσω να απαντήσω. Λοιπόν, η πρώτη ομάδα είναι ποιους ίδιους πόρου θα πρέπει να δημιουργήσουμε και ποια είναι τα προβλήματα σε σχέση με τους συγκεκριμένους ίδιους πόρου. Το πρώτο έχει να κάνει με τα κριτήρια που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να προσδιορίσουμε αυτούς τους ίδιους πόρους. Εγώ προσπάθησα στην παρουσίασή μου εν συντομία να τα παρουσιάσω και θα βρείτε και προτάσει για συγκεκριμένου ίδιου πόρου στην έκθεση του 2012 που υπέβαλα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όμω, τα κριτήρια που χρησιμοποίησα και που ανέφερα ήταν είτε μια οικονομική δραστηριότητα που μπορεί εύκολα να γίνει κατανοητή από τους Ευρωπαίους πολίτες, καθώς ε, θα είναι ένα αποτέλεσμα της εσωτερικής αγοράς ή τομείς όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ειδωθεί ότι διορθώνει το θέμα της φορολογικής αδικίας και προωθεί τη φορολογική δικαιοσύνη στα κράτη-μέλη. Δηλαδή έχουμε αυτά τα δύο κριτήρια για να προσδιορίσουμε τους ίδιους πόρου ε, και φυσικά μπορεί να έχουμε και πολλά άλλα παραδείγματα, ε, την περίπτωση του περιβάλλοντος ε, ή του συναφείς φόρους. Όμως τώρα, η του συναφης φορους ερώτηση είναι πώς θα το κάνουμε αυτό χωρίς να δημιουργήσουμε στρεβλώσεις. Δεν μπορώ να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις, αλλά θα απαντήσω σε δύο ερωτήσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι ε, δεν έχω μελετήσει την κάθε μία εις βάθος θα χρειαζόμαστε ενές βάθο μελέτη και μερικέ φορέ. δεν έχουμε και τα δεδομένα για να μελετήσουμε τον πιθανό αντίκτυπο. Όμω, το ένα είναι η σφορά της ψηφιακή ενέργεια αγοράς και υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι στρέβλωσης. Και εγώ εργάζομαι με κάποιους συναδέλφους και προσπαθώ να δω αν είναι δυνατό να σχεδιάσουμε ένα μηχανισμό που να αποφεύγει τις στρεβλώσεις. Και χωρίς να έχω μία οριστική θέση, μπορώ να σας πω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε με τη διαφάνεια. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε το χάρη που τα έσοδα ε, ουσιαστικά δημιουργούνται από τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες. Δεν υπάρχει διαφάνεια από πού προέρχονται τα έσοδα, ε, τη διαφήμιση το χάρη των ε, μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών ε, και δεν ξέρουμε τα έσοδα, δεν ξέρουμε τις πιθανές τρευλώσεις, δεν ξέρουμε πώς κατανέμονται κτλ και νομίζω ότι η κοινή ενωπημένη βάση φορολογίας εταιριών μπορεί να βοηθήσει να διορθώσουμε αυτό το πρόβλημα. Όμως δεν νομίζω ότι το, η διόρθωση αυτού του προβλήματος θα πρέπει να εξαρτάται από τη CCTB από την κοινή ενωπημένη βάση φορολογία εταιριών. Νομίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει ήδη να δράσει σε αυτό. Και μια άλλη ερώτηση έχει να κάνει με το εξής. Με την ε, ε, υπερφορολόγηση των επιχειρήσεων, ε, έναν επιπλέον φόρο στι επιχειρήσει, αν θα είχε ένα στρεβλωτικό αποτέλεσμα ή αν θα δημιουργούσε, ε, παραδείγματο χάρη, μια ανισότητα, γιατί θα είχε και διασυνορικό χαρακτήρα. Αυτός ο πρόσθετος φόρος θα ισχύει, θα εφαρμοζόταν σε όλε τι επιχειρήσει, ανεξάρτητα με το αν έχουν διασυνορική δραστηριότητα ή όχι. Αυτό που είπα, αν έχουμε τι πληροφορίε βάσει τη κοινή βάση φορολογία εταιριών, μπορούμε τότε στο επίπεδο της ε, κατανομής ε, ε, του εισοδήματος να δώσουμε ένα μέρος αυτών των εισόδων στα κράτη-μέλη και ένα άλλο μέρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα λάμβανε μόνο τα έσοδα που θα συνδέονται με τη διασυνοριακή δράση αυτών των εταιριών. Όμως ο φόρος θα φορούσε όλη την οικονομική δραστηριότητα αυτών των εταιριών. Τα έσοδα από αυτόν τον επιπρόσθετο φόρο που θα πήγαιναν για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα σχετίζονταν με τις ε, δραστηριότητες των επιχειρήσεων που καθίστανται δυνατές σε βάση της ενιαία αγορά, τη εσωτερική αγορά. Και η δεύτερη ερώτηση ήταν κυρίω ε, πολιτική και σχετίζεται με το πώ θα το υλοποιήσουμε αυτό και πώ θα πείσουμε τα κράτη-μέλη. Το πρώτο μου επιχείρημα θα ήταν είναι ότι θα έχετε ένα πιθανό βραχυπρόθεσμο πολιτικό κόστος έναντι ενός πολύ χαμηλότερου πολιτικού κόστους στο μέλλον. Γιατί δεν θα έχετε πλέον το ιδιαίτερα υψηλό κόστος συναλλαγών που έχετε στα πλαίσιο του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου και τη συζήτηση του προπολογισμού, γιατί δεν θα είχατε αυτή τη συζήτηση για το Zero Sum Game, όπως κάνετε σήμερα, ούτε θα είχατε το εσωτερικό πολιτικό κόστος που έχετε σήμερα. Είναι δύσκολο να διαπραγματευτεί κανείς το πολιτικό δημοσιονομικό οικονομικό πλαίσιο, γιατί κατόπιν εθνικέ κυβερνήσει πρέπει να πάνε και να το πουλήσουν σε εισαγωγικά εγχωρίω. Και ξέρετε το πολιτικό κόστο που πληρώνουν σε εσωτερικό επίπεδο ε, λόγω τη πρώτη που έδειξα μπορείτε να καταλάβετε. Όμως, αν πάτε στις ίδιου πόρους θα έχετε χαμηλότερο πολιτικό κόστος γιατί δεν ε, θα συνδέεται με το πόσο θα συνεισφέρει το κράτος μέλος από τον ε, εθνικό του προπολογισμό. Ε, Έχοντα περάσει τρία χρόνια στην πολιτική, γνωρίζω πόσο δύσκολο είναι να αλλάξουμε το βραχυπρόθεσμο πολιτικό κόστο για μεσοπρόθεσμο πολιτικά ωφέλη. Ξέρω ότι θα είναι κάτι δύσκολο Κατά την έποψή μου, πολιτικά πολλά θα κερδιθούν σε επίπεδο κρατών μελών και εθνικών κυβερνήσεων, όμω φυσικά υπάρχει ένα βραχυπρόθεσμο πολιτικό κόστο και είναι πιο δύσκολο να ληφθούν οι αποφάσει λόγω αυτού. Τώρα, πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτό το βραχυπρόθεσμο πολιτικό κόστος. Νομίζω πολλοί από εσά ήδη είπατε πιθανά στοιχεία της διαπραγματεύσης θα μειώσουν το πολιτικό κόστος εσωτερικά πέρα από την επιλογή που θα κάνετε σε σχέση με του ίδιου σπόρους. Όμω, αν μειώσετε τις εισφορές εκαθάρισης του εθνικού εισοδήματο ταυτόχρονα, τότε αυτό θα είναι ένα τρόπο να το πουλήσετε σε εθνικό επίπεδο αν ε, δημιουργήσετε ε, μια εναλλακτική στη φορολογική εναρμόνιση, τότε αυτό μπορεί να βοηθήσει και κάποια κρατημέλη και πάλι να το πουλήσουν. Αν χρησιμοποιήσετε κάποιου από του ίδιου πόρου για να καταπολεμήσετε την ε, φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή, αυτό μπορεί να μας σα επιτρέψει ταυτόχρονα να μειώσετε ακόμη και το ΦΠΑ. Και έτσι θα το πουλήσετε ως κάτι θετικό, κάτι που μειώνει το φορολογικό άχθος ε, στους πολίτες. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι μπορούμε να προσπαθήσουμε πολιτικά να σχεδιάσουμε μια δεσμή μέτρων, αλλά θα πρέπει να εργαστείτε σε κάθε ένα ξεχωριστό επίπεδο προκειμένου να σημειώσετε επιτυχία και όπως είπα μακροπρόθεσμα και μέσο πρόθεσμα δείχνουν ξεκάθαρα τα στοιχεία ότι αυτό θα μείωνε το πολιτικό κόστος για το κράτη-μέλη και τις, και τις εθνικές κυβερνήσεις σε ό,τι αφορά την προοπτική ανέντεξη. Εμείς σας ευχαριστούμε και τον καθηγητή Άντορ θέλω να ευχαριστήσω που βέβαια αποχώρησε αλλά ευχαριστώ την απουσία του και τον κύριο Άντορ ευχαριστώ και σας κύριε Μαδούρο και προχωρούμε τώρα στο δεύτερο σκέλος αυτής της ακρόασης ε, που είναι η φορολογική εναρμόνιση ε, και οι κινητές βάσεις, φορολογικές βάσεις Έχουμε την Εμμανουέλα Μενσάν καταρχάς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι η τομεάρχη στην γαμαδέλτα budget ε, για τον έλεγχο των ιδίων πόρων βάσει του ΦΠΑ μεταξύ άλλων. Ήρθε τον Οκτώβριο του 2003 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει εργαστεί σε διάφορες γενικές διευθύνσεις όπως μεταξύ άλλων επιχειρήσει, μεταφορά ενέργεια, οικονομικά, νομισματικά. Προηγουμένως έχει απασχοληθεί σε διάφορες ε, Ομάδε ε, προβληματισμού Think Tank, το CREDO, Research Certified Study and Monitoring of Living Standards. Έχει ε, διδακτορικό στα εφαρμοσμένα οικονομικά, είναι υπεύθυνη για την απόφαση των ιδίων πόρων σε επίπεδο της μονάδας που ηγείται και είναι και στην ομάδα εργασία για του ίδιου πόρου στο Συμβούλιο Εκ Μενσά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μου δίνει τη δυνατότητα να σας παρουσιάσω εδώ την πρότασή μας. Φυσικά θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω τη σχέση που υπάρχει με τις πολιτικές μας, ποιο είναι το σκεπτικό πίσω από αυτή την πρόταση. Χαίρομαι που βλέπω τα πράγματα θα είναι εύκολα για μένα σήμερα το πρωί, διότι οι περισσότεροι από εσάς ε, έχετε ήδη μεγάλη εξοικείωση και γνώση του φακέλου θα είναι δηλαδή πράγματα γνωστά σε εσά τα πιο πολλά που θα πω. Θα ήθελα όμως να σας δώσω και κάποιες ε, πιο λεπτομερείς εξηγήσει ε, για τον γιατί θεωρούμε ότι είναι σημαντική η μεταρρύθμιση του συστήματος. Θα ήθελα να σας εξηγήσω ότι προσπαθούμε να πετύχουμε και ίσως επίσης να κάνω μια άμεση σχέση μεταξύ των προτάσεων μας για τους ίδιους πόρους και των πολιτικών και προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με αυτή την πρόταση. Καταρχάς, θα σας δώσω κάποια βασικά μηνύματα για να σας δείξω το γιατί και το πώς ε, σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση του συστήματο των πόρων. Όπω ξέρετε, αυτή τη στιγμή έχουμε τρει ε, ίδιου πόρου οι οποίοι χρηματοδοτούν συνολικά τον προπολογισμό κατά 90%. Έχουμε του τελωνιακού δασμού. Ο παλαιότερος στασμός ε, που είχε να κάνει με τη βασική ε, δραστηριότητα της Ένωσης την εμπορική δραστηριότητα χρηματοδοτείται από τους ελληνικούς ασμούς για το στο 13%. Έπειτα έχουμε ε, τον ίδιο πόρο που βασίζεται στο ΦΠΑ, δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 70 σε συνάρτηση με την προσπάθεια εναρμόνισης και του καθεστώτος του ΦΠΑ στα κράτη-μέλη. Έχουμε εξοδηγίες που εγκρίθηκαν το 1977 για το σκοπό αυτό και έχουμε και το καθάριστο εθνικό εισόδημα. Το 1988 προτάθηκε και αρχικά υποτίθεται ότι θα δυστυχούσε σε ένα μικρό μερίδιο του ενωσιακού προπολογισμού, αλλά όπως είπατε και ορισμένοι εξημών, τώρα έχει φτάσει να χρηματοδοτεί σχεδόν το 70% του ενωσιακού προπολογισμού. Και βέβαια αυτή είναι και η δυσκολία. Όπως όλοι καταλαβαίνετε, Όλα πηγαίνουν πολύ καλά, πολύ ικανοποιητική η χρηματοδότηση του ενωσιακού προπολισμού με αυτούς τους τρεις ίδιους πόρους. Γιατί ξέρετε ότι η ισορροπία είναι ο ισοσκέλης του προπολογισμού, είναι ε, πρωταρχικός ε, κανόνας. Και τον πέτυχε αυτό ε, το σύστημα. Είχαμε τις πιστώσεις πληρωμών, μετά είχαμε τις τολωνιακούς δασμούς και το ΦΠΑ που μπορεί να κυμαίνεται ο ε, σπόρος από το ένα έτος άλλο και έπειτα έχουμε το εθνικό εισόδημα που είναι ένας εξισορροπητικός αν θέλετε ίδιο σπόρος. Ακούστηκαν κάποιες φωνές που λένε ναι μεν, αλλά γιατί ε, να μεταρρυθμίσουμε κάτι που λειτουργεί και αυτό είναι σωστό. Υπάρχει σοσκελισμένος προπολογισμό κάθε χρόνο και τα κράτη-μέλη μάλιστα κάθε χρόνο ε, με βάση το ε, ακαθάριστο εθνικό εισόδημα ε, παίρνουν πίσω ίσως κάποια χρήματα και υπάρχει αυτή η ισορροπία, αυτή η ισοσκέληση του προπολογισμού. Τελευταία προσπάθεια μεταρρύθμισης του συστήματος ήταν το 2011 το αποτέλεσμα ήταν όχι νέοι ήδη οι πόροι, αλλά η ομάδα σοφών του Μόντι που αναφέρθηκε. Η τελευταία μεταρρύθμιση ήταν πριν από 30 χρόνια. Και έχουμε αυτούς τους τρεις είδους πόρους που έχουν κριθεί επιτυχημένοι. Και αυτό εξηγεί τη δυσκολία του εγχειρήματο της μεταρρύθμισης του συστήματος. Αυτό είναι το χρονικό υπόβαθρο είναι το ιστορικό έκθεση Μόντι, τη γνωρίζετε, δεν θα σας ε, πω ε, περισσότερα. Η τελική έκθεση δημοσιοποιήθηκε το 2016 και το 2018 είχαμε την πρόταση της Κομισιόν για την τροποποίηση του συστήματος. Ποιο είναι το σκεπτικό πίσω από αυτή την πρόταση. Μπορούμε να τον δούμε από δύο διαφορετικές προοπτικές ε, το σύστημα αυτό. Ότι ήταν ένα επιτυχημένο σύστημα. Άρα, αφού λειτουργεί σωστά, γιατί να το αλλάξουμε, θα ρωτήσουν κάποιοι. Και αυτό είναι σωστό βέβαια. Το δεύτερο όμως είναι ότι ο κόσμος αλλάζει, προσπαθούμε τις δαπάνες να τις εξυγχρονίσουμε. Με τις δαπάνες ε, ε, και την προστέμενη αξία, δημόσια αγαθά, η κλιματική αλλαγή είναι μια πρόκληση σε ευρωπαϊκό και φυσικά και σε παγκόσμιο επίπεδο, εσωτερική αγορά, που ακούστηκε και πολύ σε αυτή τη συνάντηση, δαπανούστηκαν και δαπανώνται πόροι για την ε, εσωτερική αγορά. Έχει σίγουρα ένα κόστος αυτή η επιτυχία, αλλά έχει και πολλά ωφέλη και πρόσφατα δημοσιοποιήθηκαν ε, μελέτες οικονομολόγων που λένε, για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, για την περίοδο 2021-2027 έχουμε ε, υπολογίσει ένα μέσο όρο 0,9% το εθνικό καθάριστο εισόδημα Εθνικέ εισφορές δηλαδή, που δεν ξεπερνάνε το 1% επαναλαμβάνω, ούτε καν το φθάνουν. Η εσωτερική αγορά ωφελείται σε ποσοστό 6% του καθάριστου εθνικού εισοδήματος, με βάση τις μελέτες. 5% για τη Γερμανία είναι το ποσοστό, η τη Γαλλία 15% για το Λουξεμβούργο, 11% για τη Σλοβακία κτλ. κτλ. Αυτό όμως το οποίο δεν γίνεται αντιληπτό ως όφελος γιατί υπάρχουν αυτοί οι εξωτερικοί παράγοντες, θετικοί εξωτερικοί παράγοντες, ε, δεν είναι προφανές, αλλά οι πολίτες ωφελούνται καθημερινά και οι επιχειρήσεις. Αλλά στην καθαρή θέση ε, ή στις εισφορές δεν το βλέπουμε ξεκάθαρα αυτό. Και αυτός είναι και ο πρώτος λόγος που χρειάζεται μετάρρυθμιση στο σύστημα για να συνδεθεί με τον προπολογισμό και τις προτεραιότητες της Ένωσης. Υπόθηκε και σήμερα νωρίτερα. Πουθενά δεν ε, παίζει ρόλο το τμήμα των εσόδων σε καμία πλευρά του κόσμου. Δεν υπάρχει που το, τα έσοδα να μην παίζουν κανένα ρόλο. Θέλουμε να πλουστεύσουμε τους ιδίους πόρους. Μετά από 30-40 χρόνια λειτουργίας του συστήματος, φυσικά και πρέπει να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Εκπτώσεις, τα rebates. Προτείνουμε να καταργηθούν σταδιακά μέσω ενός καταποκοπήν ποσού, Uh, Ο κ. Φερνάντης ε, έκανε μια αναφορά σε αυτό το σύστημα με τις εκπτώσεις. Uh, και έχουμε επίσης και την κυκλική οικονομία και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής που είναι προτεραιότητες. Στο γράφημα αυτό, στα δεξιά βλέπετε ότι έχουμε την διαφοροποίηση. 12% περίπου με τους νέους ίδιους πόρους, άρα το μερίδιο του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος μειούται αυτή την πρόταση. Εν συντομία τώρα θα ήθελα να σας πω τι έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε και πώς συσχετίζουμε τους διάφορους στόχους ε, με τις προτεραιότητες. Έρχομαι στον ΦΠΑ, ε, τον ε, λιγότερο έτσι, θετικά ειδωμένο πόρο από τους περισσότερους. Σχετίζεται με την εσωτερική αγορά, ήταν επιτυχημένο, παρέχει σταθερό προβλέψιμο σταθερά προβλέψιμα έσοδα για τον προπολογισμό της Ένωσης και ήταν και ένας από τους πρώτους ίδιους πόρους που σχετίστηκε με τη φορολογική εναρμόνιση. Όμως, πράγματι, έχει γίνει πολύπλοκο το σύστημα του ΦΠΑ. Πώς να σας το πω, διότι ο στόχος του ήταν στο δυνατόν πιο δίκαιο ο σύστημα. σε κάποιες ομοσπονδικές χώρες η Γερμανία για παράδειγμα, ε, υπάρχει αυτή η κατανομή του ΦΠΑ, των εσόδων από το ΦΠΑ. Αλλά δεν είναι πολύπλοκοι υπολογισμοί γιατί στα διάφορα ομοσπονδιακά κρατήρια οι συντελεστέ είναι ίδιοι. Στην Ένωση τα κράτη-μέλη μπορούν, έχουν την ελευθερία να ορίσουν του συντελεστέ του, έχουμε διάφορα ε, επίπεδα, διαφορετικού φορολογικού συντελεστέ και γι' αυτό θέλουμε να μπορούμε να τον υπολογίζουμε για να έχουμε ένα ποσοστό. Και έχουμε αυτού του υπολογισμού που προκαλούν παθιασμένε συζητήσει για την πολυπλοκότητα του ΦΠΑ. Αυτό που προσπαθήσαμε λοιπόν να κάνουμε είναι να έχουμε έναν υπολογισμό της βάσης ε, του ΦΠΑ για να απλοποιήσουμε τα πράγματα ε, και ξεκινάμε με ε, τα εθνικά έσοδα και προσπαθούμε στην πρότασή μας να εξελίψουμε τον πολύπλοκο υπολογισμό των αντισταθμίσεων, των ε, διορθώσεων ε, για να είμαστε όσο δυνατόν πιο κοντά στην οδηγία ΦΠΑ, όπως θα εφαρμοζόταν η οδηγία ΦΠΑ πλήρως, χωρίς εξαιρέσεις και παρακλήσεις. Έτσι λοιπόν, απλώς ε, φορολογούμε τα έσοδα και έχουμε μια ουδετερότητα. Εδώ, δεν ξέρω αν μπορείτε να διαβάσετε τη διαφάνεια. Έχετε δύο γραφήματα και βλέπετε τα βήματα των υπολογισμών μας. Αν δείτε το πρώτο δεξιά, εδώ συγκρίνουμε τα ακαθάριστα έσοδα, όπως τα λαμβάνουν στους εθνικούς προϋπολογισμούς στα κράτη-μέλη, ε, συγγνώμη, τα, τα καθάριστα έσοδα και τα καθαρά έσοδα, όπως λαμβάνονται από τα κράτη-μέλη και την Κομισιόν. Βλέπω ότι ουσιαστικά δεν υπάρχουν διαφορές. Αυτό σημαίνει ότι αν ξεφορτωθείτε τις διορθώσεις, δεν υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά και αυτό είναι τεράστια πλούστευση για μας και για τα κράτη-μέλη. Το δεύτερο γράφημα αριστερά συγκρίνουμε την ενδιάμεση βάση με την τελική βάση. Ε, Αυτή την ορολογία χρησιμοποιούμε, αλλά τα κράτη-μέλη τα γνωρίζουν αυτά, γιατί τα χρησιμοποιούν στα στοιχεία που δίνουν στην Κομισιόν. Και εδώ, να σας πω ποιο είναι το μέγεθος, έχουμε περίπου 25 αποζημιώσεις που είναι ε, η κυρία δουλειά ελέγχου της Κομισιόν. Επίσης, έχουμε περιορισμένες διαφορές. Βλέπετε καταρχήν ότι αν εξαλείψουμε τις αντισταθμίσεις και τις διορθώσεις δεν πλήττεται ε, η ολότητα, η κεραιότητα της βάσης, αλλά είναι πολύ πιο απλή η έλεγχη. Και αυτό είναι σημαντικό. Δεύτερον, έχουμε πολύ καλά νέα ότι η φορολογική εναρμόνιση στο ΦΠΑ είναι ψηλή. Και αυτά είναι καλά τα νέα και ίσως σχετίζεται με την επιτυχία του ΦΠΑ. Και τρίτον, μέσω της απλούστευσης που προτείνουμε, μπορούμε να διατηρήσουμε την ακαιρεότητα της σύνδεσης των ιδίων πόρων με το ΦΠΑ να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για το πώς ε, λειτουργεί. Όταν η Κομισιόν ε, ελέγχει τα κράτη-μέλη, το ΦΠΑ, έχουμε κοινή αποστολή γύρω στα ταξούτ και μπάτζετ, γιατί έχουμε απλή εφαρμογή της οδηγίας για το ΦΠΑ. Απλώς αυτό για να σας δείξω ε, ποιο είναι το θέμα της φορολογικής ενερμόνησης και της CCTB. Συγγνώμη, και της ιστορικής αγοράς, δεν μιλήτρια. Τώρα, η CCTB, Κοινή Ενωπημένη Βάση Φρολογίας Επιχειρήσεων, ε, ήταν ε, πρότασή μας ε, το 2018. Δεν υπήρχε όρεξη από τα κράτη-μέλη, θα ήταν λοιπόν κάπως πρόημο να το έχουμε. Η λογική ήταν σύμφωνα με αυτά που ακούσαμε στο πρώτο πάνελ, δηλαδή ότι ουσιαστικά ε, βασιζόμαστε στην πρόταση που ε, ξαναπαρουσιάστηκε από την Κομισιόν το 2016 και είχαμε ε, ουσιαστικά έναν επιμερισμό των κερδών στα κράτη-μέλη και ποιο θα ήταν το η λογική αν δούμε τις μεγάλες εταιρείε τότε ε, ουσιαστικά ένα μεγάλο μέρος ε, των κερδών είναι εκτός της εσωτερικής αγοράς ε, σε άλλα κράτη-μέλη. Έτσι λοιπόν αυτό ήταν το λογικό για να σχετίσουμε τους ίδιους σπόρους με την ιστορική αγορά σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση των επιχειρήσεων. Κατόπιν έχουμε δύο πράσινους ίδιους σπόρους τη συνεισφορά από τα πλαστικά. Και αυτό συνδέεται με τις προτεραιότητες τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει δεσμευτικούς στόχους για την ανακύκλωση για τα πλαστικά και άλλα υλικά. Εδώ θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε ένα συντελεστή για ε, τα απόβλητα πλαστικών ε, που ε, παράγουν τα κράτη-μέλη και ένα θετικό αντίκτυπο, ένα θετικό αποτέλεσμα είναι ότι θα δημιουργήσουμε ένα κίνητρο για τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν την ανακύκλωση και υπάρχει ουσιαστικά ένα είδο εναρμολόγηση των μεθοδολογιών που, χρησιμοποιούνται από τα κράτη-μέλη και τώρα συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη για να βελτιώσουμε την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων. Και επίση, ε, πολλή δουλειά γίνεται και από του συναδέλφου τη Eurostat για να δώσουν ε, κατεύθυνση και υποστήριξη στα κράτη-μέλη για να βελτιώσουν τα στατιστικά στήματα για πιθανού ίδιου πόρου σε αυτό. Και κάτι τελευταίο, το σύστημα εκπορία ε, εκπομπών που αναφέρθηκε πολλάκι εδώ. Και αυτό είναι μια ε, επιτυχία στην ε, νέα πολιτική, δηλαδή για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική απειλή, την κλιματική αλλαγή, συγγνώμη, και ουσιαστικά να συστορικοποιήσουμε το κόστος ε, των εκπομπών του αερίου του θερμοκηπίου. Τώρα, έχουμε μία τιμή για τον άνθρακα, και μία ή δύο πλατφόρμες δημοπρασιών που λειτουργούν. Έτσι λοιπόν δεν χρειάζεται να σας πείσω γιατί κάναμε την πρόταση για να έχουμε 20% των εσόδων από τις δημοπρασίες ε, που θα πηγαίνουν στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Είναι πάρα πολύ εύκολο για μας να το θέσουμε σε αυτοερμογή, δεδομένου ότι υπάρχει η πλατφόρμα αυτή δημοπρασίας και ουσιαστικά τα έσοδα από τις σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιστρέφουν στον εθνικό προϋπολογισμό. Επομένως και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι μέρος της προσθέμενης αξίας της ευρωπαϊκής πολιτικής. Αυτή είναι η λογική για τους ίδιους πόρους, για κάθε ίδιο πόρο. Ε, ε, of comparison. Να περάσουμε στη σύγκριση. Το πρώτο γράφημα δεξιά. Δεν θα έλεγα ότι αφορά το μέγεθος, μην επικεντρώνεστε στο μέγεθος ε, του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, αλλά να πω ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός δεν θα πρέπει να ειδωθεί μεμονωμένα. Γιατί πάντοτε υπάρχει ένα σύνδεσμος. Ξέρετε, όταν εργαζόμουν στην ΕΚΦΗΝ, ε, ε, λέγανε ότι δεν υπάρχουν σύνορε της οικονομίας, Είναι αλήθεια, αλλά ο ευρωπαϊκό προπολογισμό δεν μπορεί να ειδωθεί ε, απομονωμένο από του πολίτε και του εθνικού προπολογισμού. Αν ε, συγκρίνουμε τα συστήματά μα, ε, βλέπετε ότι έχουμε περίπου παρόμοια δομή μεταξύ των εθνικών κρατών και ομοσπονδιακών συστημάτων. Δεν είναι ομοσπονδιακό σύστημα η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά βλέπετε πώ δουλεύει. Έχουμε ε, εθνικέ εισφορέ και φεύρει περιβαλλοντικό φόρο, εταιρικό φόρο, από αυτά προέρχεται η χρηματοδότηση και φόρο κατανάλωσης. Υπάρχουν ε, ε λοιπόν ε, κοινά στοιχεία μεταξύ εθνικού και ευρωπαϊκού επίπεδου και αυτό θέλουμε να δείξουμε με το γράφημα στα αριστερά. Βλέπετε με την διαφοροποίηση των ιδίων πόρων έχουμε μεγαλύτερη φορολογική συνοχή μεταξύ ευρωπαϊκού προπολογισμού και των εθνικών προπολογισμών. Όμως ε, δεν είναι μόνο θέμα δομής αυτό, θέλουμε να συνάδουμε και με τις εθνικές οικονομικές εξελίξεις, να ε, συνάδουμε με τις ε, ευρωπαϊκές οικονομικές πολιτικές. Ε, ξέρετε ότι κάποιες οικονομίες πάνε πιο γρήγορα, παραδείγματο χάρη, στη μετάβαση σε καθαρές τεχνολογίες. Δηλαδή, αν έχουμε ε, διαφοροποίηση στους ίδιους πόρους, ε, ουσιαστικά ε, τα έσοδα του ευρωπαϊκού προπολογισμού θα τα συνδέσουμε και με άλλες παραμέτρους που συνδέονται με τις εθνικές οικονομίες. Και εδώ θέλω κάτι σημαντικό να πω, γιατί εξακολουθεί να υπάρχει το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα και έχουμε νέους ίδιου ε, και αν διατηρήσουμε τη ΦΠΑ δεν σημαίνει ότι θα ξεφορτωθούμε το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα, το αντίθετο γιατί ήδη οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα έλεγα ότι είναι κάτι που έχει φτιαχτεί καλά. Δηλαδή είναι σε ισορροπία ο προπολογισμό σε σχέση με το καθάριστο εθνικό εισόδημα. Έτσι λοιπόν διατηρούμε αυτό το επαγγελματικό τείχο ε, του καθάριστο εθνικού εισοδήματο ε, και αν κάνουμε υπολογισμού προ τα πίσω και έχουμε και το καλάθι των ε, νέων πόρων με το κόκκινο, με την κόκκινη γραμμούλα το βλέπετε αυτό, θα δείτε ότι στην πραγματικότητα αν είχαμε διαφοροποίηση των ιδίων πόρων το 2005 τότε το μερίδιο του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος θα ήταν χαμηλότερο. Αλλά θα βλέπετε ότι θα ήταν πιο κυκλικό το καθαριστό εθνικό εισόδημα, γιατί η διαφοροποίηση των ίδιων πόρων βασίζεται στην κυκλικότητα των εθνικών οικονομιών, της προτεραιότητας, των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό σημαίνει ότι προωθεί, η μεγιστοποίηση την, ε, το μηχανισμό της ε, αλληλεγγύης και επιμερισμού ε, του συστήματος. Δηλαδή διατηρούμε την ακαιρεότητα της λειτουργίας του συστήματος. Και θέλω να κλείσω. Δεν προτείνουμε εδώ μία επανάσταση, απλώς έναν εξυγχρονισμό έναν εξυγχρονισμό προκειμένου ε, ουσιαστικά τα έσοδα να συνεισφέρουν στη χάραξη των ευρωπαϊκών πολιτικών, να συνεισφέρουν στον προπολογισμό και να είναι πιο συναφή με τις εθνικές οικονομίες. Βεβαίως, ε, άκουσα ε, σήμερα το πρωί ε, πολλά σχόλια. Η Κομισιόν είναι ανοιχτή και πρόθυμη να εξετάσει νέες προτάσεις που δίνουν στο τραπέζι. Αλλά εγώ πιστεύω ότι μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι αν έχουμε κάποιους ένα-δύο νέους ίδιους πόρους θα είναι ένα μεγάλο βήμα. Γιατί η τελευταία μεταρρύθμιση που είχαμε ήταν το 1998. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Πίτερ Πάλους, ο οποίος είναι επικεφαλής του Τμήματος Οικονομικής Πολιτικής στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι μέλος της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής καθώς επίσης και του Euro Working Group. Ασχολείται με ζητήματα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, οικονομικών υποθέσεων, φορολόγησης, τελωνίων καθώς επίσης και συντονισμού κρατικών ενισχύσεων είναι υπηρεσιακό αναπληρωτή υπουργό στο Υπουργείο Οικονομικών τη Σλοβακία. Συμμετέχει στι συνεδριάσει του Eurogroup και παίρνει επίση πολύ συχνά το λόγο, καθώ επίση και δημοσιεύει αρκετά άρθρα στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Κύριε Πάλου, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητοί καλεσμένοι, σας ευχαριστώ καταρχάς κύριε Πρόεδρε για τα πολύ θετικά σας λόγια. Θα ήθελα να διαρθρώσω την παρουσίασή μου σε δύο βασικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα θα επικεντρωθεί στην θέση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ποια είναι η στάση της Σλοβακικής Δημοκρατίας και η προσωπική μου στάση όσον αφορά του ιδίους πόρους, καθώς επίσης και το ζήτημα της εναρμόνιση τη φορολογική πολιτική. Η δεύτερη δενότητα θα επικεντρωθεί σε τέσσερα βασικά μηνύματα, τα οποία κατά την άποψή μου είναι θεμελιώδου σημασία αν θέλουμε να επιτύχει το όλο εγχείρημα, ξεκινώντας καταρχά με την θέση του Συμβουλίου. Όπως ενδεχομένω γνωρίζετε, το Συμβούλιο είναι αρκετά διχασμένο όσον αφορά το ζήτημα των ιδίων πόρων. Έχουμε περίπου 7 κράτη-μέλη, τα οποία είναι διαλλακτικά και ανοιχτά στην ιδέα της συζήτησης νέων πιθανών ιδίων πόρων. Υπάρχουν άλλα κράτη-μέλη τα οποία σιγά-σιγά κινούνται προς την ομάδα αυτή, προς την κατεύθυνση αυτή. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι η πλειονότητα των κρατών μελών στο Συμβούλιο είναι σαφώς κατά της ε, δημιουργίας νέων ιδίων πόρων και προσπαθούν και μάλλον προτιμούν τις συνεισφορές μέσω του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος. Τώρα, η φορολογική εναρμόνιση. Πώς αντιμετωπίζεται αυτή από το Συμβούλιο. Ως προς αυτό, καταρχάς, θα πρέπει να καταλάβουμε τι εννοούμε ή πώς ορίζουμε την έννοια της φορολογικής εναρμόνισης. Αν η βασική ιδέα πίσω από την έννοια αυτή είναι να τροποποιήσουμε το εφιστάμενο σύστημα ψηφοφορίας στο Συμβούλιο και να περάσουμε από την ομοφωνία στην ειδική, πλειοψηφία, στην ειδική ψηφοφορία, ειδική πλειοψηφία, τότε τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερα θετικά στο Συμβούλιο. Υπάρχουν ε, πολλές χώρες που εξακολουθούν και συντάσσονται περισσότερο με την ομοφωνία και χώρες οι οποίες ανησυχούν για το ότι ενδεχομένως να αρχίσει να κινδυνεύει η έννοια της φορολογικής κυριαρχίας. Και σε αυτό συμβάλλουν επίσης και κάποια άλλη φόβη όσον αφορά την έννοια της, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως πολιτική ένωση. Ξέρω πάντως ότι η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Φοντελάιεν, προβλέπει μία μελλοντική διαβούλευση, διάσκεψη για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα διαρκέσει δύο χρόνια και θα ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της επερχόμενης Γαλλικής Προεδρίας. Πρέπει να δούμε πώς θα κινηθούν τα πράγματα τα επόμενα αυτά δύο χρόνια, αλλά θα πρέπει καταρχάς να πετύχουμε μια συμφωνία για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πάντως, απευθυνόμενο σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρέπει να σας πω ότι Όντα στο κτίριο Μπερλεμόν τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είδα ότι το βασικό μήνυμα είναι μια Ευρωπαϊκή Ένωση που καταβάλει προσπάθειε προκειμένου να πετύχει περισσότερου και ανώτερου στόχου. Θα ήθελα να επανέλθω τώρα στο ζήτημα της φορολογικής εναρμόνισης. Αν ουσιαστικά εννοούμε ότι σε κάποιους ε, τομείς ε, θα μπορούσαμε να προβλέψουμε φορολογία εκεί πέρα που δεν προβλέπεται. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν ήδη κάποιες προτάσεις που συζητώνται στο Συμβούλιο και πρέπει να σας πω ότι στον τελευταίο πολιτικό κύκλο, τα τελευταία δηλαδή τέσσερα χρόνια, καταφέραμε να συμφωνήσουμε για πάνω από 30 ψηφια... Ε, νομοθετικές προτάσεις στον τομέα της φορολογίας και αυτό αποτελεί θεωρώ τεράστιο επίτευγμα. Η πρόοδος που έχουμε σημειώσει στον τομέα αυτή είναι πολύ υψηλότερη και πολύ σημαντικότερη από τα επιτεύγματα των τελευταίων 50 χρόνων. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ πέρα τα πράγματα κινούνται θετικά και η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει τελικά ότι ακόμα και η διαδικασία ψηφοφορία μέσω ομοφωνία στο Συμβούλιο για προλογικά ζητήματα λειτουργεί θετικά στην πράξη. Δεύτερον, όσον αφορά τώρα την θέση που έχει οθετήσει η δική μου χώρα, η Σλοβακία. Όπως σας είπα υπάρχουν 7 κρατημέλη τα οποία είναι διαλλακτικά στην όλη συζήτηση για τους ιδίους πόρους, ιδίως στον τομέα του περιβάλλοντος. Και εντασσόμαστε και εμείς σε αυτά τα 7 κρατη Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να καταρτήσουμε νέους ιδίους πόρους, επειδή συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει ανάγκη διαφοροποίησης και ανάγκη σταθεροποίησης των πόρων του ενουσιακού προπολογισμού. Νομίζω ότι το εξήγησε πολύ καλά ο καθηγητής Άντορ πριν από λίγο. Δεν θα ήθελα λοιπόν να επανέλθω στο σημείο αυτό. Και βλέπουμε ότι ιδίω στον τομέα του περιβάλλοντος ισχύει αυτό. Στον τομέα του περιβάλλοντος θα έλεγα ότι όλο και περισσότερο βλέπουμε να υπάρχει μια αναδυόμενη συνένεση όλων πλέον των κρατών μελών αλλά και στην ίδια την κοινωνία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι κάτι επιτέλους πρέπει να κάνουμε, ότι πρέπει να αναλάβουμε δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος. Θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε ενώπιόν μας μια μοναδική ευκαιρία να αξιοποιήσουμε το φορολογικό σύστημα για να πετύχουμε τους περιβαλλοντικούς μας στόχους. Και θα έλεγα ότι αυτός είναι και ο πιο αποτελεσματικό τρόπος για να τροποποιήσουμε τη συμπεριφορά των πολιτών, τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Ας μην χάσουμε λοιπόν τη χρυσή αυτή ευκαιρία που έχουμε μπροστά μας, ας την αξιοποιήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Εμμανιουέλ μας έδωσε κάποια παραδείγματα, αναφέρθηκε σε κάποιες συγκεκριμένε ιδέες με τις οποίες συμφωνώ. Θα πρέπει για παράδειγμα να έχουμε μια συνεισφορά η οποία να προκύπτει από τις μη ανακυκλωμένες πλαστικές συσκευασίε. Θα μπορούσαμε επίσης να έχουμε και ένα διασνοριακό φόρο άνθρακα ή ακόμα και μία επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών. Όλα αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν τμήμα της ε, τελικής δέσμης που θα αποφασίσουμε για τους ίδιους πόρους. Όσον αφορά τώρα την φορολογική εναρμόνιση, ε, η δική μου χώρα και εγώ ίδιος έχουμε μία επιφυλακτική προσέγγιση. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε το σύστημα ψηφοφορίας όσον αφορά τα φορολογικά ζητήματα και ξέρουμε ότι κάθε φορά που μιλάμε για φόρους έχουμε ιτημένου και νικητέ. Αυτό ισχύει και για τα κράτη-μέλη. Αν αλλάξουμε λοιπόν τον τρόπο ψηφοφορία για τα ε, φορολογικά ζητήματα, ενδεχομένως ε, τα μικρά κράτη-μέλη να βρίσκονται πραγματικά στο έλεος ε, των αποφάσεων των μεγάλων κρατών μελών. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να καλύψουμε ενδεχομένω με τι φορολογίε κάποιου τομεί τη οικονομία που δεν καλύπτονται. Είμαστε ανοιχτοί στο να γίνει μια τέτοια συζήτηση και σα έδωσα ήδη κάποια παραδείγματα όσον αφορά το περιβάλλον. Παρ' όλα αυτά, εν γέννη, νομίζω ότι ο τομέας τη έμεση φορολογίας θα μπορούσε να αξιοποιηθεί περισσότερο για την ε, δημιουργία ευρωπαϊκών φόρων που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στον κοινοτικό προπολογισμό. Θα μπορούσα ω προ αυτόν να σα δώσω κάποια ακόμα παραδείγματα. Αναφέρθηκαν κάποιοι στον φόρο επιχρηματοστοτικών συναλλαγών. Θα μπορούσαμε εδώ να συμπεριλάβουμε και του ψηφιακού φόρου, τον φόρο γκάφα για παράδειγμα. Θα μπορούσαμε να έχουμε και άλλες μορφές έμεσης ε, φορολογίας στο πλαίσιο τη ε, ενιαία αγορά και θα μπορούσε και αυτό να συνεισφέρει στον κοινοτικό προπολογισμό. Τώρα, ποια είναι η προσωπική μου άποψη. Εγώ θεωρώ ότι ε, νέοι ναι, ήδη πόροι θα ήταν επωφελεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι πεπισμένο γι' αυτό. Θα έλεγα μάλιστα ότι ε, ο σημαντικότερος λόγος για κάτι τέτοιο και νομίζω ότι αναφέρθηκε πολλές φορές αυτό σήμερα είναι το ότι στα πλαίσια του ενωσιακού προπολογισμού χρησιμοποιούμε μόνο την πτυχή των δαπανών. Δεν χρησιμοποιούμε καθόλου την πτυχή των εσόδων του ενωσιακού προπολογισμού προκειμένου να διαμορφώσουμε την συμπεριφορά των πολιτών μας, προκειμένου να διαμορφώσουμε την πολιτική που ακολουθούν οι επιχειρήσεις μας. Και θεωρούμε ότι θεωρώ ότι εδώ χάνουμε μια πολύ σημαντική ευκαιρία. Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα, το φόρο για την αεροναυτιλία, τις αεροπορικές μεταφορές. Θα μπορούσαμε και στις μεταφορές αυτές να έχουμε έναν πανευρωπαϊκό ενωσιακό φόρο που θα συνεισφέρει στο κοινοτικό προπολογισμό. Νομίζω ότι πρωταρχικός μας στόχος στην περίπτωση ενό τέτοιου φόρου θα ήταν να πείσουμε τους πολίτες να χρησιμοποιήσουν πιο φιλοπεριβαλλοντικούς τρόπους μεταφορών και να μειωθεί κατά αυτόν τον τρόπο το επίπεδο εκπομπών διεξιδίου του άνθρακα, που τους άλλω αυτό αποτελεί προτεραιότητά μας. Θα ήταν καλό επίσης να μπορούσαμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο να έχουμε έναν συλλογικό ομαδοποιημένο φόρο με τον οποίο να συμφωνούν όμως όλες οι χώρες. Η ε, Σλοβακία, για παράδειγμα, δεν θα μπορούσε να συμφωνήσει από μόνη της για έναν φόρο επί των αεροπορικών μεταφορών, αν αυτός ο φόρος δεν, δεν τον συμμερίζονται και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Δεν νομίζω ότι είναι ένας φόρος που θα μπορούσε μονομένα να εγκριθεί από τα κράτη-μέλη. Θα μπορούσαμε και άλλου φόρους να έχουμε στον τομέα της αεροναυτιλία. Υπάρχουν νησιωτικές χώρες όπως η Μάλτα ή η Κύπρος που εξαρτώνται όπως καταλαβαίνετε πολύ περισσότερο από τι αεροπορικέ μεταφορές. Νομίζω λοιπόν ότι και στην περίπτωση αυτή θα μπορούσε να υπάρχει, όπως σας είπα, αυτή η αμοιβαία συλλογική προσέγγιση, ένας επιμερισμός του φορολογικού, ε, της φορολογικής εισφοράς που θα μπορούσε να προκύψει προκειμένου να μην επιβαρύνονται με μονομένες χώρες που εξαρτώνται πάρα πολύ από τις ε, αεροπορικές μεταφορές. Υπάρχουν επίσης άλλες χώρες που θέλουν να διατηρήσουν την υφιστάμενη κατάσταση, το status quo. Και θεωρούν επίσης ότι μπορεί να προκύψει ακόμα και ένα άφελος από τον φορολογικό ανταγωνισμό. Εμείς δεν χρησιμοποιούμε όμως ως Σλοβακία αυτό το φορολογικό ανταγωνισμό ή δεν προκύπτει για μας κάποιο φορολογικό πλεονέκτημα, θέλετε, από αυτό το ανταγωνισμό. Τώρα να περάσω στο δεύτερο σκέλος της ε, παρέμβασής μου, να αναφερθώ σε τέσσερα βασικά μηνύματα, όπως σας είπα. το οποίο νομίζω ότι θα μας βοηθήσουν να ολοκληρώσουμε το όλο αυτό το εγχείρημα με επιτυχία. Και εδώ θα μπορούσε να θέσει κανείς και κάποια ερωτήματα. Θα πρέπει καταρχάς να έχουμε νέους ιδιοσπόρους. Θεωρώ πως ναι. Πρέπει να έχουμε νέους γνήσιους ιδιοσπόρους στον νοσιακό προπολογισμό. Σαφώς ναι. Δεύτερον, θα πρέπει να έχουμε φορολογική εναρμόνιση, να βασιστούμε σε αυτήν. Θεωρώ πως όχι. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο αν δεν δώσουμε πιο έντονο πολιτικό χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρώ ότι μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια θα ήταν δύσκολο να καταλήξουμε σε πλήρη φορολογική εναρμόνιση. Και Προκειμένου να πετύχουμε αυτή την εναρμόνιση θα πρέπει να γίνουν και πολλές άλλες οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Τρίτον, θα πρέπει να προκύψουν συνέργειες, αυτό το βλέπουμε και στον τίτλο της σημερινής ακρόασης. Συνέργειες ανάμεσα στις δύο αυτές πτυχές, τα δύο αυτά ζητήματα. Πάλι αρνητική απάντησή μου. Το να διασυνδέσουμε τη φορολογική εναρμόνιση και τους ιδίους πόρους σε μια ενιαία ενότητα θα μπορούσε να είναι ακόμα και αντιπαραγωγικό και θα μπορούσε να λειτουργήσει και εις βάρος της εξέβρεσης νέων ιδίων πόρων. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους νέους ιδίους πόρους ως πρόσχημα για να προχωρήσουμε τελικά σε μια φορολογική εναρμόνιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος και εξίσου σημαντικό, η άποψη των Ευρωπαίων πολιτών για όλα αυτά. Το ζήτημα δηλαδή της νομιμοποίησης. Ας μην ξεχνάμε ποτέ την άποψη του μέσου Ευρωπαίου πολίτη. Διότι βλέπουμε ότι αναδύονται διάφορα λαϊκιστικά κινήματα παντού στην Ευρώπη, τα οποία θα χρησιμοποιήσουν τις εξελίξεις αυτές και θα πούνε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή στυλιτεύει την φορολογική κυριαρχία, την εθνική φορολογική κυριαρχία των κρατών μελών. Εν κατακλείδη να πω ότι δεν θα πρέπει να συγχαίουμε ιδίου πόρου και φορολογική εναρμόνιση και αν θέλουμε πραγματικά να στεφτεί με επιτυχία το όλο αυτό εγχείρημα, α μην συνδέουμε του ιδίου πόρου με το συνολικό όγκο του τελικού ενωσιακού προπολογισμού. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να μειώσουμε σε καμία περίπτωση το επίπεδο του ενωσιακού προπολογισμού, ούτε θα πρέπει οι ίδιοι πόροι να λειτουργήσουν ει βάρο των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν αυτοί οι νέοι ήδη πόροι, θα πρέπει να εξευρεθούν, αλλά θα πρέπει να υποκαταστήσουν άλλες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι ε, θα πρέπει να προβλέψουμε ένα κατάλληλο επίπεδο προπολογισμού, στον ενωσιακό προπολογισμό, που ακόμα όμω και το κατάλληλο αυτό επίπεδο πάλι θα συναντήσουμε αρκετού περιορισμού. Τα χρήματα ουσιαστικά ποτέ δεν θα φτάνουν. Γι' αυτό νομίζω θα πρέπει να αρχίσουμε να αξιοποιούμε λίγο περισσότερο την πτυχή των εσόδων στον ενωσιακό προπολογισμό. Σα ευχαριστώ πολύ. Το λόγο οι συνάδελφοι για σχόλια, ερωτήσει. Κύριε Ανδρέα, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση χωρίς μικρόφωνο. Δεν ακούγεται από τους διερμηνείς. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Your mic, your mic, your mic. Sorry. Το μικρόφωνο σας. Α, συγγνώμη, μίλαγα χωρίς να ξέρω ότι είχα κλειστό το μικρόφωνο τόση ώρα. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω κάτι για το φόρμα προσαρμογή ε, στα σύνορα, για τον άνθρακα. Όχι τόσο όσον αφορά το περιεχόμενο, αλλά το χρονοδιάγραμμα. Διότι οι πληροφορίες μου λένε ότι η πρόταση θα, κατέ... θα είναι έτοιμη το 2021. Τότε θα κατατεθεί. Τώρα όμως εμείς έχουμε ήδη ξεκινήσει να το συζητάμε. Και η πρόεδρος της Κομισιόν, κυρία Φοντρελάιεν, ξέφρασε ισχυρά επιχειρήματα και έκανε δηλώσεις και στην κοινή γνώμη και το κόμμα της στην Γερμανία ήδη, ε, το, στρέφεται ενάντια αλλά το 2021 είμαστε πολύ μακριά είναι αυτή η ημερομηνία. θέλουμε πρόοδο στη συζήτηση και αν θέλουμε ένα σενάριο κοφόρο πρέπει να κινηθούμε πολύ πιο γρήγορα και όχι να ξεκινήσουμε με την κατάθεση μιας πρότασης το 2021. Η συγκεκριμένη ερώτηση που σας ε, υποβάλλω είναι είναι έτσι το χρονοδιάγραμμα. Θα καταθέσετε κάποια πρόταση το 2021 ή νωρίτερα κάτι συγκεκριμένο. Γιατί εμείς θα θέλαμε να συνδεθεί με τις διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ένα γενικό μήνυμα. Διερμηνία έχουμε μέχρι τις 12 και 10. Μπορούμε να συνεχίσουμε, απλά δεν θα έχουμε διερμηνία μετά τις 11 και 10, ή 12 και 10. Κυρία Αγιέ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τους δύο ομιλητές μας, Μεσόν και Πάλους. Μία παρατήρηση και ερώτηση την κυρία Μεσόν και μια ερώτηση για τον κύριο Πάλους. Η παρατήρηση είναι η εξής. Μιλήσατε για τα ωφέλη της εσωτερικής αγοράς για τα κρατημέλη. Λυπούμε, αν κατάλαβα τουλάχιστον καλά αυτά εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, είναι δύσκολο να έχουμε στρατηγικού ε, χαρακτήρα πληροφορίες από την Κομισιόν, που μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμες παρόλα αυτά, παραδείγματο χάρη για τα ωφέλη, ε, για τα κρατημέλη από την εσωτερική αγορά. Αυτά τα είχαμε, παραδείγματο χάρη, τα στοιχεία πέρυσι, στο τέλος του χρόνου. Σε μια μεγάλη γερμανική εφημερίδα έγιναν κάποια σχόλια και ενευρίασε ο κύριο Έτιγκερ και έτσι πήραμε εμεί αυτέ τι πληροφορίε που ήταν πραγματικά πάρα πολύ σημαντικέ γιατί ουσιαστικά ε, βοηθούν είναι θετικά αυτά. Είναι επιχείρηματα υπέρ μας. Εσείς έχετε αυτές τις πληροφορίες, ε, στατιστικά στοιχεία ή και εντυπώσεις και ε, κοινή γνώμης. Θα ήταν καλύτερα να τα ε, διανέμετε σε εμά περισσότερο, να μας τα διαβιβάζετε, για να έχουμε και συγκλίνουσες θέσεις. Αυτή είναι η παρατήρηση. Ερώτηση. Μιλήσατε για την απλούστευση του ΦΠΑ ως ίδιου πόρου. Η Κομισιόν τι θα κάνει μετά την ε, ευρεία άποψη που κυκλοφορεί στο Συμβούλιο υπέρ της κατάργησης του ΦΠΑ ως ίδιου πόρου. Δεν μας ανησυχεί ως ευρωβουλευτές η θέση αυτή. Γιατί είναι και εκτιμένα αυτά που δεν πρέπει να τα βάλουμε, να τα θέσουμε από αμφισβήτηση. Και αν όμως περάσει κάτι τέτοιο, αν καταργηθεί ο ΦΠΑ, έχετε κάποια αναλλακτική. Και στον κύριο Πάλους. Γνωρίζετε τα γρανάζια, το μηχανισμό εκ των έσω. για το βάσιμο του να προχωρήσουμε με μια μεταρρύθμιση του συστήματος ιδιοπόρων στο Συμβούλιο. Πώς μπορείτε να ε, πείσετε τους, ε, τους Συμβούλου που δεν συμφωνούν ή τι επιχείρηματα μπορείτε να μας δώσετε εμά για να πείσουμε τους εκπροσώπους του Συμβουλίου επί της ουσίας και σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Φερνάντες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα στενοχωρήσω την συνεισηγήτρια. Μη μας πείτε τι επιχειρήματα θέλετε να χρησιμοποιήσουμε πέρα Συμβούλιο, γιατί ακούει το Συμβούλιο και θα αλλάξει η επιχειρηματολογία. Ε, εντάξει, πλάκα έκανα. Φυσικά και μπορείτε να πείτε. Ε, το λέω έτσι για να έχουμε μια ωραία διάθεση αυτή τη συζήτηση. Συμφωνώ με τη συνεισηγητριά μου. Για το ΦΠΑ. Πώς και υπάρχουν κρατημέλη που θέλουν την κατάργηση. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Ο ΦΠΑ είναι ευρωπαϊκός πόρος που είναι σημαντικός για την εσωτερική αγορά. Βασίζεται στην ε, εσωτερική αγορά. και συνεισφέρει στην καταπολέμηση της ε, απάτης της φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής. Επομένως δεν καταλαβαίνω το λόγο για τον οποίο τα κράτη-μέλη ζητούν την κατάργησή του. Γιατί αυτό σημαίνει ότι είναι υπέρ της φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής και απάτης. Τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Κάτι ακόμη. Μια αντίφαση ακόμη που διαπιστώνουμε τα κράτη-μέλη θέλουν να διατηρηθούν εκπτώσεις και τα αντισταθμίσματα και οι αντισταθμίσεις επί αντισταθμίσεων. Μα αυτό δεν δημιουργεί μεγαλύτερη διαφάνεια. Μια ακόμη ερώτηση, έτσι, συνιστά και κάποια είδους πρόκληση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπεραμείνεται των ιδιών πόρων. Υπεραμείνεται των ιδιών πόρων που Θέλουμε κι εμείς. Και αν το κάνει, δεν το βλέπουμε στην πρόταση τόσο πολύ. Θέλει να είναι στο πλευρό μας η Κομισιόν. Έχει τη φιλοδοξία, φιλοδοξία. Τις μην μιλάμε για φιλοδοξίες. Ας μιλήσουμε για τις ελάχιστες ανάγκες, τα στοιχειώδη. Και για τους δυο σας ένα ερώτημα. Χρονοδιάγραμμα. Ετέθηκε από προλαλήσαντες. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι συζητήσει επειδή ακριβώ υπάρχει ανάγκη ομοφωνία στο Συμβούλιο, τριβούμε γενικώ, καθυστερούμε στο Συμβούλιο. Αλλά το 2021 πρέπει να ξεκινήσει το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο. Στη δική μας τη θέση είμαστε ξεκάθαροι. Ζητούμε μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων. Νέους ίδιους πόρους. Αλλιώς δεν θα έχουμε νέο πι δελτα πι. Θα βιαστεί το Συμβούλιο, θα βοηθήσει, θα σπρώξει λίγο την Κομισιόν. Ευχαριστώ. Merci, Madame Κυρία Μάρκες. Ευχαριστώ και εγώ για τις δύο παρουσιάσεις, ε, δυστυχώς. Την πρώτη, από την πρώτη δεν τα κατάλαβα όλα. Βέβαια, το χρόνο του χρονοδιαγράμματος ε, σχετίζεται με την ερώτηση που έθεσα στο προηγούμενο πάνελ. Όμως, η πολύ συγκεκριμένη ερώτησή μου είναι η εξή. Ε, χτες η Επίτροπος Γιώχανσεν εδώ μας είπε σε σχέση με τις ίδιους σπόρους, ότι η Επιτροπή έχει πολλές ιδέες. Αυτή τα είπα εγώ. Έτσι λοιπόν η ερώτησή μου είναι ε, είστε στο τμήμα ιδίων πόρων. Σε ποιου ιδίου πόρους, θέλω να ρωτήσω, εργάζεται η Κομισιόν, για ποιου ίδιου πόρου εργάζεται για να παρουσιάσει νομοθετικέ προτάσει. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις αυτές, λέει η κυρία Μανσάν. Συγγνώμη αν δεν τα καταλάβατε όλα από την παρουσίασή μου. γιατί είναι πάντοτε μια πρόκληση. Και φυσικά εγώ σας έδειξα ότι το σύστημα θα μπορούσε να είναι απλό, αλλά μερικές φορές ε, είναι πρόκληση να μπορεί κάποιος να παρουσιάσει απλά στοιχεία για τους ίδιους πόρους. Λοιπόν, να αναφερθώ στα διάφορα σχόλια. Λοιπόν, για το Border Carbon Adjustment. Εργάζονται οι άλλες γαμαδέλτα σε αυτό. Ε, Το ανέφερε και η κυρία Φοντερ Λάιεν στο Green Deal και στις κατευθυντήριες γραμμές. Ε, έτσι λοιπόν, είναι νωρίς να πούμε τώρα που ακριβώς ε, θα μπει ο φόρο, γιατί δεν έχουν γίνει ακόμα μελέτε αντικτύπου, τεχνική δουλειά από την Κομισιόν κτλ. Είναι κάπω νωρί λοιπόν για, πας, για να πούμε ποια μορφή θα πάρει. Ξέρω ότι περισσότερο το χρονοδιάγραμμα αφορούσε η ερώτησή σας. Τώρα, ότι έχουμε καθυστερήσει, ναι, ο στόχος είναι να έχουμε συμφωνία το συντομότερο. και κατά τη διάρκεια του έτους και το συζητήσει για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο ε, ίσως θα μπορέσουμε να το δούμε, όμως ε, μέχρι τώρα δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε επί του Border Carbon Adjustment. Ε, φυσικά, όπως αναφέρθηκε σήμερα το πρωί, αν θα συνδεθεί και με το σύστημα εμπορίας εκπομπών θα το δούμε. Αν ήμασταν επιτυχείς ε, με αυτό, τότε αυτό θα μπορούσε να είναι κάτι που θα το σκεφτούμε. Θα επανέλθω στους σπόρους ΦΠΑ. Ναι, συνειδητοποιούμε ποια είναι η θέση της πλειοψηφίας των κρατών μελών. Δεν ξέρω αν είμαι αισιόδοξη. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι όταν εργαζόμαστε επί των ιδιών πόρων. Όμως αυτό που καταλάβω από τις, κατασ... σε τεχνικό επίπεδο είναι η πρώτη επιλογή της πλειονότητας κρατών μελών να καταργηθεί ο ΦΠΑ. Όμως ε, κάποιοι εκφράσαν ε, και ανοιχτέ θέσεις σε μία-δύο μεθόδους απλουστευσής που προτείναμε. Δεν ε, θα μπω τώρα στις τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά είχαμε μία παρουσίαση το Μάιο. Που, πώς να το πω, δεν έτυχε θετικής ανταπόκρισης από κάποια κράτη-μέλη. Και για να λάβουμε υπόψη τις ανησυχίες κάποιων κρατών μελών, προτείναμε άλλη μέθοδο πλούστευσης. Πού βρισκόμαστε τώρα. Είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι. ότι μία από τις δύο αυτές εναλλακτικέ θα μπορούσε να ειδωθεί θετικά από όλα τα κράτη. Ξέρουμε ότι για κάποια κρατημέλη αυτό το τελικό γραμμή και για το Συμβούλιο φαντάζομαι ότι είναι ένα, ένα θέμα που θα είναι αντικείμενο των διαπραγματεύσεων. Δεν έχουμε στρατηγική αναδίπλωση αυτή τη στιγμή. Θεωρούμε ότι είναι ιστορικός πόρος και όπως σας είπα και σας έδειξα, επίσης αποτελεί επιτυχία και προς τις δύο κατευθύνσεις. Δηλαδή, θεσπίσαμε αυτό τον ιδιοφόρο βάση της εσωτερικής αγοράς, αλλά επειδή πρόκειται για ιδιοπόρο, συνεισέφερε και στην επιτυχία της φορολογικής εναρμόνισης. Επομένω, ε, γνωρίζουμε ότι με τη μεθοδολογία που προτείναμε και τις θέσεις των κρατών μελών ε, θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε. όχι για την εσωτερική αγορά. Κοιτάξτε, και εγώ δυσκολεύομαι να εκφραστώ. Μας ξεπερνά μερικέ φορές. Λοιπόν, φυσικά ω Κομισιόν, στο μέτρο που μπορούμε, υποστηρίζουμε όλε τις τεχνικέ συζητήσει. Είμαστε διαθέσιμοι, εκτός των τελευταίων μηνών, παίξαμε το ρόλο αυτό κατόπιν αιτήματος ε, της τεχνικής ομάδας όπου συμμετέχουμε. Είμαστε λοιπόν ανοιχτοί να συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε αυτό το ρόλο και στο μέλλον. Είπατε, κυρία Χάν, ότι έχουμε πολλές ε, ιδέες ε, και σίγουρα οι ομάδες μου εργάζονται για κάθε πιθανή εναλλακτική, ανεξαρτήτως πολιτικού προσανατολισμού. Και αυτό εξηγεί γιατί πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για να μπορούμε να έχουμε επιτελέσματα σε τεχνικό επίπεδο. Και φυσικά εξετάσαμε όλες τις ιδέες που αναφέρθηκαν στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας, της επέκτασης του ETS, του Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών και του Μηχανισμού Προσαρμογής στα σύνορα, αλλά ακούσαμε και το θέμα του ψηφιακού φόρου, του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και όλα αυτά ε, τα έχουμε ακούσει και έχουμε εργαστεί επί αυτών σε τεχνικό επίπεδο. Αυτά ήθελα να πω. Κύριε Σπάλους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία αυτή που μου δίνεται για να ευχαριστήσω τους συνεισηγητές Χολμάιερ και Φερνάντες για την εργασία που έχουν επιτελέσει όσον αφορά το σημαντικότατο αυτό ζήτημα, το οποίο νομίζω ότι είναι σημαντικό για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να κάνω κάποιες σύντομες παρατηρήσεις. Όσον αφορά το μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα. Ακούσαμε την άποψη του Κοινοβουλίου ότι θα πρέπει να καταρτιστεί και να ελοπιθεί το συντομότερο δυνατό και είπαμε ότι υπάρχουν όλο και περισσότερες χώρες στο Συμβούλιο που τάσσονται υπέρ του μηχανισμού αυτού, άρα καλό θα να κινηθούμε στο δυνατό γρηγορότερα. Τώρα, όσον αφορά τη συνεισφορά βάση του φόρου προστιθέμενης αξίας, από ό,τι φαίνεται, Ορισμένα κράτη-μέλη θεωρούν ακόμα ότι το όλο σύστημα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο και θα χρειαζόντουσαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και απευθύνομαι στη Μανουέλ περισσότερε εξηγήσει. Το πιο σημαντικό θέμα είναι αυτό που έθεσε όμως η Βαλερή. Δηλαδή, πώς θα καταφέρουμε τελικά να πείσουμε τα κράτη-μέλη εκείνα, τα οποία απέχουν πάρα πολύ από τη δική σας τη θέση, να εξευρεθούν δηλαδή νέοι ή ήδη πόροι. Ο καθηγητής Μαντούρο νομίζω ότι το ανέφερε αυτό, όταν μίλησε για το πολιτικό κόστος νομίζω ότι θα πρέπει αυτό να το έχουμε κατά νου. Δηλαδή, τι συμβαίνει σε επίπεδο εθνικών κυβερνήσεων. Και έπειτα, ποια είναι η μεγαλύτερη ανησυχία που έχουν οι εθνικές αυτές κυβερνήσεις. Το ότι ενδεχομένω να απολέσουν τον έλεγχο της φορολογικής τους πολιτικής, τον έλεγχο του μεγέθους του νοσιακού προπολογισμού και όλα τα παρεπόμενα. Γνωρίζουμε τις ανησυχίες αυτές, ωστόσο εγώ θα ήθελα να ξέρω το ακόλουθο και το θέτω αυτό σαν ανοιχτό ερώτημα και προς εσάς. Προς τα μέλη δηλαδή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν τελικά ο απότερος στόχος μας για τους νέους ιδίους πόρους είναι να καταφέρουμε να σταθεροποιήσουμε τον ενωσιακό προπολογισμό αν πραγματικά θέλουμε να διαφοροποιήσουμε τις πηγές του ενουσιακού προπολογισμού, αν θέλουμε τελικά να διαμορφώσουμε καλύτερα την πτυχή των εσόδων των κοινοτικών πολιτικών ή μήπως κρύβονται άλλες προθέσεις πίσω από την ιδέα αυτήν. Μήπως πίσω από τους νέους ίδιους πόρους θέλουμε να αυξήσουμε τον όγκο του προπολογισμού και να οδηγηθούμε τελικά σε φορολογική εναρμόνιση. Αυτό είναι λοιπόν το ερώτημά μου. Αν η απάντησή σας είναι ότι τελικά πίσω από την ιδέα των νέων ιδίων πόρων θέλουμε τελικά να ενισχύσουμε την πτυχή των εσόδων και να διαμορφώσουμε καλύτερε νοσιακέ πολιτικέ, τότε νομίζω ότι το εγχείρημα αυτό θα στεφτεί με επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρο. Ολοκληρώνεται κατά αυτόν τον τρόπο η πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συνεδρίασή μα. Να ευχαριστήσω καταρχά του εμπειρογνώμονε μα για τι εξαιρετικέ παρουσιάσει του για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους και να ευχαριστήσω βέβαια και τα μέλη της Επιτροπής μας για την δική τους τη συμβολή. Νομίζω ότι καταφέραμε να ακούσουμε πολλά ενδιαφέροντα επικοδομητικά επιχειρήματα προς όλες τις κατευθύνσεις και ελπίζω ότι βάση της συζήτησης αυτής θα μπορέσουμε να έχουμε μια πολύ πιο επικοδομητική συζήτηση εν συνεχεία για τον ουσιακό προπολογισμό. Σας ευχαριστώ πολύ.